Αγαπητοί συνάδελφοι, οι συντονιστές αποφάσισαν να επιτρέψουν το ακόλουθο και θα ήθελα να σας ζητήσω αυτή τη στιγμή να κάνετε ησυχία. Πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα με την εργασία της Επιτροπής μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά σημεία στη μερίσια διάταξη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο στον εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, μιας οργάνωσης από την Πολωνία για μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Good morning everybody. My name is Małgorzata. Καλημέρα σας. Γκούρσκα ονομάζομαι. Είμαι από την Πολωνική Οργάνωση για την Προστασία των Πτηνών είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Είμαι και εγώ αναφέρουσα και μαζί με τους συναδέλφους μου από άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις της Πολωνίας υποβάλαμε μία αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά έναν δρόμο ο οποίος θα σχεδιαζόταν στην Πολωνία και ουσιαστικά θα έβλαπτε ε, προστατευόμενες περιοχές από το Natura 2000 στην Ανατολική Πολωνία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και τα μέλη και άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μαζί καταφέραμε να τροποποιήσουμε την απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης και να σώσουμε περιοχές όπως αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, την κοιλάδα στην Ανατολική Πολωνία. Σώθηκε λοιπόν η περιοχή αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνετε για να σας ευχαριστήσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Την υποστήριξή σας μας επέτρεψε να σώσουμε το πολύτιμο αυτό μέρο στην Πολωνία και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να σώσουμε και άλλα τέτοια πολύτιμα μέρη σε άλλε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ε, Απρίλιο το Ίδρυμα Goldman των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να δώσει ένα οικολογικό βραβείο Νόμπελ, μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, για την εκστρατεία μας αυτή. Πήγα λοιπόν σαν Φραντζίσκο και είχα την τιμή να παραλάβω το βραβείο αυτό και για άλλη μια φορά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους γιατί συνεβάλλετε κι εσείς στο να μας δοθεί το βραβείο αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε για την ακοίνωση αυτή, λέει η Πρόεδρος. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Μέρκη έχει ζητήσει τον λόγο για κάτι διαδικαστικό όμω. Ναι, ναι, ναι. Στην ημερήσια διάταξη θα ήθελα να αφαιρθώ και θα ήθελα και εγώ να κάνω μια προσωπική δήλωση και θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Μπορώ να κάνω αυτή τη δήλωση, σας παρακαλώ πολύ, και μπορώ να σχολιάσω και την ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη τώρα, στις παρατηρήσεις που έχουμε. Πρόεδρος, ε, αναφέρεστε στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Κοιτάξτε, αν θέλετε να πάρετε το λόγο για σημείο της ημερήσιας διάταξης, τότε θα το κάνετε αυτό, τότε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όχι, λοιπόν. Θα ήθελα να πω ότι όντως θέλω να συζητήσω για την ημερήσια διάταξη. και συγκεκριμένα το ζήτημα έχει να κάνει με την καμπανία και θα ήθελα να κάνω και μία δήλωση προσωπική και να συμπεριληφθεί αυτό και στη μερίσια διάταξη. Μπορώ να κάνω κάποια σχόλια για τη μερίσια διάταξη τώρα. Πρόεδρος, κυρία Μέρκης, κοιτάξτε, η καμπανία δεν συμπεριλαμβάνεται στη μερίσια διάταξη. Κοιτάτε ενδεχομένω τη μερίσια διάταξη της συνάντησης των συντονιστών. Εκεί συζητήθηκε Η ημερήσια διάταξη τη συνεδρίασή μα όμως τώρα τη Επιτροπής δεν προβλέπει σημείο για την καμπανία. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ήδη καθυστερήσει από χθε. 10, 11, 12 είναι τα σημεία τα οποία δεν προλάβαμε να εξετάσουμε χθε. Κυρία Μέρκη, μπορείτε να μου πείτε πότε θα καταφέρω να κάνω αυτή την προσωπική μου δήλωση που θέλω να κάνω. Δεν κατάλαβα το αίτημά σας. Τι θέλετε, να πάρετε το λόγο για την καπανία. Σας είπα δεν περιλαμβάνετε στη μερίσια διάταξη. Κυρία Μέρκης, όχι. Δύο πράγματα θέλω να κάνω. Πρώτον, να μιλήσω για την ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα για την καμπανία και επιπλέον κάτι εντελώ διαφορετικό, να κάνω μια προσωπική δήλωση. Αυτό είπα. Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια στιγμή στην ημερήσια διάταξη την απαραίτητο χρόνο ώστε να κάνω τη δήλωσή μου αυτή. David Law κοιτάει εδώ πέρα τον κανονισμό, επομένως θα μου πει τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα επιπλέον σημείο στη μερίσια διάταξη. Στο διάμεσο διάστημα με την δική σας σύμφωνη γνώμη θα ήθελα να προχωρήσουμε τη μερίσια διάταξη. αναφορά 1403 κάθτος 2007 της κυρίας Ντομπρίνκα Παυλόβα. Δεν είναι παρούσα η αναφέρουσα. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάδελφός μου, κυρία Σταβίνοβα, δεν είναι εδώ. Γιωχάννα Ίνστραγκ ονομάζομαι και θα αναφερθώ και στις τρεις αναφορές που έχετε στα σημεία 10, 11 και 13, αν δεν κάνω λάθος. Παύλοβα, Ντέσμοντ Φιτζέραλτ και Παυλίνα Ράτκοβα. Όλες αυτές τις αναφορές θα ήθελα να τις εξετάσω μαζί γιατί αναφέρονται σε πάνω κάτω ίδια ζητήματα. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνείτε? Ναι, λέει ο Πρόεδρος. Οι αναφορές έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία στη Βουλγαρία. Ιδίω τα παιδιά αυτά τα οποία βρίσκονται σε ορφανοτροφία και ιδρύματα τη Βουλγαρία, ζήτημα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο ντοκιμαντέρ του BBC το Σεπτέμβριο του 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλέ φορέ έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή των Αναφορών για το ζήτημα αυτό και σε έχουμε δώσει πολλέ γραπτέ δηλώσει και ανακοινώσει συνεχίσαμε να εργαζόμαστε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και έχουμε έρθει σε επαφή με τις αρχές της Ρουμανίας προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνική προστασία των παιδιών με αναπηρίες. Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η βασική ευθύνη για την προστασία των παιδιών και την ενσωμάτωση των παιδιών παραμένει βασική αρμοδιότητα ακόμα των κρατών μελών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία είναι, τα οποία είναι πλήρως αρμόδια για την προάσπιση των ε, δικαιωμάτων αυτών στα πλαίσια των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λοιπόν άμεση αρμοδιότητα για να εξετάσει, για να επέμβει στην κατάσταση των ε, παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα, ούτε μπορούμε να επέμβουμε στο σύστημα το οποίο προβλέπεται από τη ρουμανική κυβέρνηση για την βοήθεια και τη φροντίδα των παιδιών, όπως αναφέρεται άλλωστε στην αναφορά της κυρίας Ράτκοβα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτουν αναφορές και είμαστε δεσμεύοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τα παιδιά στα ιδρύματα αυτά και τις οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία στη Βουλγαρία. Στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας περιγράψαμε τις γενικότερες δράσεις που έχουν αναλυφθεί. Αναφερθήκαμε στις ε, μελέτες που έχουν γίνει και έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκαμε στις δονισμό πολιτικών και σε ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Θα θέλαμε επίσης να αναφερθούμε στην ad hoc επιτροπή που δημιουργήθηκε από τον Επίτροπο Σπίτλα το Φεβρουάριο του 2009, η οποία επέβαλε και μία έκθεση το Σεπτέμβριο του 2009 Πρόκειται για μια έκθεση η οποία αναφέρεται στην υποστήριξη κατά την μετάβαση από τα ιδρύματα προς οργανισμούς που βασίζονται στην κοινότητα για τα παιδιά τα οποία έχουν αναπηρίες. Γίνονται στην έκθεση αυτή διάφορες συστάσεις. Μία από, αυτή, μία από αυτές αναφέρεται στην επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες θα πρέπει να σημειώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Αν περάσουμε τώρα στι συγκεκριμένε δράσει που έχουν αναλυφθεί σε σχέση με τη Βουλγαρία, πρέπει να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα συνεχή σταθερό διάλογο για τη μεταρρύθμιση των Ιδρυμάτων για τα παιδιά με αναπηρίε και έχουμε υποστηρίξει τι προσπάθειε τη Βουλγαρία προκειμένου να καταλήξει σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική μεταρρυθμίσεων και πάρα πολλέ από τις βουλγαρικές πρωτοβουλίες τις έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενε ανακοινώσει μας. Βλέπετε ότι μετά από προσεκτική ανάλυση της κατάστασης στη χώρα αυτή, η βουλγαρική κυβέρνηση τελικά πρόσφατα έλαβε κάποια μέτρα προκειμένου να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις και έχει κλείσει κάποια μεγάλα ιδρύματα όπως το Μοχιλίνο αν επικεντρωθούμε στις πιο πρόσφατες δράσεις της Βουλγαρίας που ήρθαν μετά από δική μας γραπτή απάντηση, βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον ένα σχέδιο δράσης της Βουλγαρίας το οποίο καλύπτει μια περίοδο 10 με 15 ετή, πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουν, πώς μπορούν αυτοί να βοηθήσουν πολύ περισσότερο τα παιδιά τα οποία φεύγουν από τα ιδρύματα και πηγαίνουν σε άλλους οργανισμούς και έχει εξεταστεί το πρόγραμμα αυτό από το Συμβούλιο Υπουργών τη ε, Βουλγαρίας. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε ένα άλλο μέσο για να υποστηρίξει τη χώρα. Τα χρηματοδοτικά μέσα, τα διαφορετικά ταμεία συγκεκριμένα έχουν χρησιμοποιηθεί. Και πέρα από αυτά που σα είπαμε στο παρελθόν, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε μία πρόσφατη πρωτοβουλία που λέγεται «Let us not leave a single child behind», α μην ξεχάσουμε κανένα παιδί πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και η ΑΤΧΟΚ Επιτροπή του Επιτρόπου Σπίτλα. Ξεκίνησε το 2010 η πρωτοβουλία αυτή, βρίσκεται στα πρώτα της στάδια προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δούνε ποιε είναι οι ανάγκε των παιδιών που βρίσκονται ακόμα σε ιδρύματα στην Βουλγαρία. Αυτό γίνεται από μια πολυεπιστημονική ομάδα 250 ιατρών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματιών στην Βουλγαρία. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέοι οργανισμοί, σαν οικογένειε που θα μπορούσαν ουσιαστικά να φιλοξενήσουν τα παιδιά αυτά. Και η προσπάθεια αυτή, όπω σα είπα, χρηματοδοτείται από τα διευθυντικά ταμεία. Επίση, στα πλαίσια τη νέα στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μέσα Νοεμβρίου, θα είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε τη στρατηγική αυτή και να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να βοηθήσουμε την μετάβαση από τα ιδρύματα σε οργανισμούς οι οποίοι οργανώνονται από τοπικές κοινότητες. Τώρα για το Μογγυλίνο είπαμε ότι εξετάζουμε την κατάσταση αυτή από το 2007. Το ίδρυμα αυτό έχει κλείσει πλέον. Την 1η Οκτωβρίου του 2009 έκλεισε συγκεκριμένα και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί, τα 75 παιδιά που ήταν εκεί και που είδατε και στο ντοκιμαντέρ του BBC, εξετάστηκαν από επιτροπή της UNICEF Ήρθαν επίσης σε επαφή με τους γονείς, τους ρώτησαν αν θέλουν να ξεκινήσουν τουλάχιστον μια νέα σχέση με τα παιδιά τους και τα παιδιά αυτά τα περισσότερα πήγανε σε κάποιες νέες μικρές δομές υποδοχής, σαν μικρές οικογένειες όπου κάθε μία φιλοξενεί 6 με 8 παιδιά. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι αναφορές αυτές μετά την απάντηση που και Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να κλείσουν. Chiede la parola sul, sul punto. Θέλει κανείς το λόγο για αυτό το σημείο. Όχι. Perfetto, quindi io ringrazio. Ε, ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή και αφήνουμε ανοιχτές τις τρεις αναφορές. Quindi, no, pensavo fosse... Mi chiedo scusa. Ε, Α, ζητώ συγγνώμη, η πρόταση ήταν να κλείσουμε τις τρει αναφορέ. Ωραία. Εντάξει. Εξαντλήσαμε τα σημεία της χθεσινής ημερήσιας διάταξης. Πάμε στη σημερινή. Τελειώσαμε με τους συντονιστές όπου συζητήσαμε τα διάφορα σημεία τα οποία θα επαναλάβω σύντομα. Η κυρία Παλιαδέλη παρουσίασε ένα αίτημα για μια έκτακτη συνεδρίαση της ε, διάσκεψης των Προέδρων με το Σώμα των Επιτρόπων όπου η κυρία Παλιαδέλη με εκπροσώπησε. Σε αυτήν τη συνεδρίαση η συνάδελφος Παλιαδέλη είχε ζητήσει το λόγο και γραπτά αλλά και σηκώνοντα το χέρι της για να παρέμβει σχετικά με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας και που αφορούσε στο θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα. Δεν της δόθηκε ο λόγος χωρίς καμία αιτιολόγηση και αποφασίσαμε να στείλουμε μία επιστολή στον πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων για να διεκδικήσουμε την ισότιμη μεταχείριση της Επιτροπής μας με τις υπόλοιπες Επιτροπές. Για το θέμα της διερευνητικής ε, αποστολής στην Καμπανία, βάσει του άρθρου 202 ζητήθηκε να παρουσιαστεί μία έκθεση για την κακή εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας στη διαχείριση των απορριμμάτων και αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσει λοιπόν η σχετική διαδικασία. Τώρα για το σημείο το σχετικό με την επίσκεψη τον Δεκέμβριο στο Κοινοβούλιο του Εδιμβούργου Περιμένουμε ένα αναλυτικότερο πρόγραμμα από τη Γραμματεία. Οι συντονιστές πάντως ε, Πέτρε, έδωσαν την, το OK για την επίσκεψη στη Σκωτία. Σημείο 3. Αναφορές για το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Ρουμανία αποφασίσαμε να κλείσουμε όλες τις αναφορές όλων των Ρουμάνων πολιτών να αφήσουμε ανοιχτές εκείνες των ενοικιαστών και να περιμένουμε την απάντηση από τον Ρουμάνο πρόεδρο. Θα ζητηθεί απάντηση λοιπόν σχετικά. Τώρα, για το σημείο το σχετικό με τη γενική ακρόαση. Συγγνώμη, συγγνώμη. Η 665-2006 του κυρίου Παραδιάς θα διαβιβαστεί στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στις αντιπροσωπίες όπως αποφάσισαν δηλαδή οι συντονιστές. Για τη γενική ακρόαση αποφασίστηκε να αναβληθεί το σημείο αυτό για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών διότι θελήσαμε να έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία. Επίσης και, το λέει, και η Λέιντε Κώστας έχει αναβληθεί διότι Έχουμε νέα στοιχεία για την εφαρμογή της Λέιντε Κώστας στην Ισπανία. Το έχουμε στα αγγλικά το έγγραφο. Δεν είχαν το χρόνο να το μελετήσουν. Θα μοιραστεί μετά από τη μετάφρασή του το κείμενο σε όλους τους συναδέλφους και θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Για την 473 κάθετος 8 του κυρίου Κλάιν που συζητήσαμε πρόσφατα και που αποφασίστηκε να παρουσιάσουμε μία ερώτηση στην Ολομέλεια διότι δεν μας απάντησε ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Δέλη, οπότε συντάξαμε μία ερώτηση η οποία εγκρίθηκε και θα παρουσιαστεί στο όνομα της Επιτροπής μας είπαμε να δώσουμε συνέχεια στην έκθεση Equitable Life στην Επιτροπή και να τη συζητήσουμε στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Επίσης προχωρήσαμε και το θέμα των μη αναφορών, των non-petition που επιβαρύνουν τη δουλειά της Επιτροπής μας και μετά από πολλά αιτήματά μας η Γενική Διεύθυνση Προεδρίας είπε ότι θα προχωρήσει σε ένα φιλτράρισμα των μη αναφορών, διότι τώρα έχουν και περισσότερο προσωπικό και θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή μας μόνο εκείνες που μπορεί να θεωρηθούν αναφορές. Και στην επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε τη διατύπωση μιας λειτουργικής πρότασης από την Επιτροπή μας. Επίσης εγκρίναμε και το χρονοδιάγραμμα του 2011 της Επιτροπής μας. Η συνάδελφος Μέρτσης θέλει το λόγο, για, η οποία θέλει να παρέμβει για προσωπικούς λόγους. Όχι. Δεν θέλω να παρέμβω για προσωπικούς λόγους για αυτό το θέμα. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στην ημερήσια διάταξη και μετά να κάνω προσωπική τοποθέτηση. Έχω μια ερώτηση για την πρόταση προετοιμασίας εκπόνησης έκθεσης για την Ολομέλεια. Θα μπορούσατε σε λεπτομέρεια να μας πείτε τι προτείνουν οι συντονιστές ή τι αποφάσισαν οι συντονιστές και ποιος θα ήταν ο ενδεχόμενο τίτλος της ε, προτινόμενης έκθεσης. Και στη συνέχεια θα κάνω την προσωπική μου δήλωση, αν μου επιτρέπετε. Ho letto quello che è stato Εγώ διάβασα, αυτό το οποίο αποφάσισαν οι συντονιστές. Και ο τίτλος της έκθεσης που προτείνεται ποιος είναι. Πώς θα φτάσει στην Ολομέλεια, ποια θα είναι η μορφή και πώς θα λέγεται αυτό το πράγμα. Διότι αρχικά ακούσαμε ότι θα πάει στην Ολομέλεια υπό το πλαίσιο ότι η Ιταλία είναι παράδειγμα ε, περιφερειών που έχουν ε, προβλήματα με τη διαχείριση των αποβλήτων. Θα συζητηθεί όμως η έκθεση στην ε, Ολομέλεια και θα δοθούν παραδείγματα και άλλων περιοχών και περιφερειών που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα πώς έχει ο τίτλος αυτής της έκθεσης. Έτσι όπως το είπα πριν. Οι συντονιστές και η Επιτροπή αποφάσισαν να πάει στην Ολομέλεια μία έκθεση η οποία θα εξετάζει το θέμα της κακής διαχείρισης και μία ορθής εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό βάσει των αναφορών που έχουμε λάβει στην Επιτροπή μας. Και βάσει αυτού να κάνετε τις παρατηρήσεις σας αγαπητοί συνάδελφε. Κυρία Πρόεδρε, ε, θα πάει στην Ολομέλη αυτή η έκθεση αναφέροντας ε, την Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ιρλανδία. Όλες τις χώρες. Λοιπόν, μην ξεκινήσουμε εδώ τώρα μια, έναν διάλογο, μια αντιπαράθεση. Λοιπόν, αν έχετε παρατηρήσεις πείτε τες και μετά να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Κυρία Πρόεδρε, δεν κάνω αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Το μόνο που σας ζητώ είναι να μου διευκρινίσετε τον τίτλο. Μπορείτε να μου διαβάσετε σας παρακαλώ τον τίτλο της εκθέσεως που θα πάει στην Ολομέλεια. Πώς θα επιγράφετε cattiva o non corretta Μη εφαρμογή των κοινοτικών νομοθεσιών στη διαχείριση των απορριμμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα να προτείνω τότε να προσθεθεί αυτό που αποφασίστηκε κατά την ψηφοφορία αρχικά, να προσθεθεί λέγω Ιταλία για να διευκρινίσουμε ότι είναι πρόβλημα σε ορισμένες περιφέρειες αυτό. Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Ιρλανδία. Συνάδελφοι Τουργάη, σου δίνω το λόγο, αλλά μην ξεκινήσουμε συζήτηση, πρέπει να κλείνει το σημείο. Θέλω. Θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα στην κυρία Μέρκης που δεν ήταν στους συντονιστές. Αποφασίστηκε στους συντονιστές. Στην αρχή είχαμε λάβει υπόψη τον τίτλο που εσείς προτείνατε. Εμείς λοιπόν στους συντονιστές συμφωνήσαμε με την αλλαγή του τίτλου και υποστηρίχθηκε και από τον δικό σας συντονιστή, τον κύριο Μπουστινάρου, δηλαδή της Σοσιαλιστικής Ομάδας, ε, η αλλαγή του τίτλου του τίτλου δηλαδή όπως τον ανέφερε η Πρόεδρος. Και επειδή η πλειοψηφία ήταν το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές για να αλλάξει αυτός ο τίτλος, άλλαξε. Τροποποιήθηκε ο τίτλος και άλλαξε. Θα πιστεύω ότι στην ομάδα σας θα έπρεπε να το είχατε ήδη συζητήσει για να μην υπάρχει αυτή η διαφορά αποφασίστηκε πλειοψηφικά η αλλαγή του τίτλου. Συμμετείχε και ο συντονιστής της ομάδας σας. Then, uh, may I... Ε, τότε ε, το γνωρίζω και σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση ε, του σημείου αυτού. ωστόσο, θα επιθυμούσα πάρα πολύ, καθώς η πρόσφατη κατάσταση στην Καμπανία δείχνει ότι είναι πήγουσα θα παρακαλούσα να γίνουν αναφορέ, Εντάξει, α μην γίνουν αναφορέ σε άλλε χώρε, αλλά να γίνει αναφορά στην Ιταλία. Γιατί αυτό δεν προτάθηκε στου συντονιστέ, λοιπόν, να βάλουμε κυρίω ιδίω η Ιταλία, ω παράδειγμα για να συζητήσει την Ολομέλεια. Αυτό κάπω μπορεί να συζητηθεί. Ε, questa è una proposta che può essere formulata attraverso il coordinatore a questo punto il gruppo dei Λοιπόν, ήταν μια πρόταση που θα έπρεπε να είχε εκφράσει ο συντονιστής. Οι συντονιστές τώρα αποφάσισαν και αυτό αποτελεί πλέον σημείο αναφορά. Λοιπόν, ο συντονιστή σα, όταν σε, στην άλλη συνεδρία, σε μια άλλη συνεδρία συντονιστών, μπορεί να κάνει τι παρατηρήσει του. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει. Λοιπόν, αν θέλετε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση, πρώτα ζήτησε το λόγο ο συνάδελφο Βίλεν και μετά η κυρία Ούκεν. Λοιπόν, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Φλιαρούμε μισή ώρα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω όλους ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκατοντάδες επίγοντα προβλήματα. Και τι δείχνει η δική μου εμπειρία εδώ και λίγες μέρες το βλέπω, αλλά ε, ε, ξαφνικά εμφανίζονται μεμονωμένοι συνάδελφοι με αγαπημένα τους θέματα και καμιά φορά και κομματική πολιτική. Έχουμε ένα κανόνα εδώ πέρα στην Επιτροπή μας, ότι αποφασίζουν κάτι οι συντονιστές και προσπαθούμε να... Ε, πώς να το πω, να μην επιφορτίζουμε την Επιτροπή μας με άχρηστη ε, Εάν θέλει κάποιο να προσβάλλει τι αποφάσει των συντονιστών, μπορεί να ζητήσει ψηφοφορία. Ο κάθε συνάδελφο. Αλλά όχι και σε κάθε συνεδρίαση. Αν θέλετε επίσημη ψηφοφορία να γίνει την άλλη φορά. Προ το παρόν η απόφαση των συντονιστών έχει έτσι και δεν χρειάζεται να τη συζητάμε τώρα εμεί εδώ. Just... Η κυρία Άουκεν, θα ήθελα μόνο να πω ότι για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργάζομαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άλλα αποφασίζουμε ομόφωνα για μια έκθεση που είναι και σημαντική και έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από μια αποστολή που μετέβηκε και ξαφνικά αγνοείται πλήρως και καταργείται αυτή η απόφαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλεύουμε με αυτές τις συνθήκες. Συμφωνώ απολύτως. Την άλλη φορά να ψηφίσουμε επισήμω ή να κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ έχασα στους συντονιστέ. Γιατί ε, φυσικά και αυτό το θέμα ε, αντικρούει τα όσα αποφασίσαμε όταν ψηφίσαμε για την έκθεση. Λοιπόν, είναι εξαίρεση. Είναι η πέμπτη φορά που παίρνετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια ε, της περασμένης εβδομάδας είδαμε να οξύνεται και να ξεσπάει νέα κρίση ε, στην υπόθεση των αποβλήτων και της διαχείρισης του στην Καμπανία. Αυτή είναι ακριβώς η έκθεση που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Διαπιστώνω, κυρία Πρόεδρε, ότι εσείς κάνατε μια δήλωση για εγκαστρίμηθους, λέτε, ευρωβουλευτές. Και ε, μέλη, λέτε, της Επιτροπής Αναφορών που χειραγωγούνται από Ιταλούς ε, βουλευτές. Θα ήθελα να αποκρούσω σφοδρότατα αυτή τη δήλωση και θα ήθελα να σέβεστε παρακαλώ το Κοινοβούλιο και να διατηρείτε τη ε, ουδετερότητα και την αμεροληψία που έχει να κάνει με τη θέση της Προέδρου. Ευχαριστώ. Ε, ε, Συνάδελφε Άουκεν, Λοιπόν, στα πρακτικά δεν διαφαίνεται τίποτα που να αμφισβητεί την αντικειμενικότητα της Προεδρίας, διότι αλλιώς αν συνεχίσουμε τη συζήτηση θα διατρέξω τον κίνδυνο να είμαι υποκειμενική λόγω και της εγκύτητας του προβλήματος το οποίο αναφέρεστε. Ο κ. Μακμέλα δεν είμαι σίγουρος ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το τι αποφάσισαν οι συντονιστέ. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έθεσε ο κύριο Παραδιά και άλλοι για τι ιδιοκτησίε και την επιστροφή, ε, υποτίθεται ε, ότι θα ρωτηθούν οι αντίστοιχε αντιπροσωπείε. Κυρία Πρόεδρε, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει κλείσει αυτή η αναφορά, σα παρακαλώ. Το επιβεβαιώνετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λό τι λέει. Η κυρία Ντεμπρούν για αυτό το θέμα, όχι για το προηγούμενο. Ε, εσείς λέτε ότι θεωρείτε αυτό που είπε για την αμεροληψία η κυρία Μέρκης ε, ανέφερε την απόφαση. Ε, αναφερόταν μάλλον στην απόφαση, όχι, αναφερόταν στη δήλωση. Γιατί εγώ συγκλονίστηκα, σοκαρίστηκα όταν είδα τη μετάφραση των όσων είπατε, ότι είναι εγκαστρίμηθο κάποιο μέλος της Επιτροπής μας. Τι είναι αυτό. Αυτό πραγματικά ε, αμφισβητεί την αμεροληψία. Και δεν είναι ευπρεπές να χρησιμοποιεί κανείς τέτοια γλώσσα για ένα μέλος της Επιτροπής μας. Προσβάλλει και θίγει και την αξιοπρέπεια και των μελών και της Επιτροπής του σύνολου. Ε, σύμφωνο Αν είχαμε δηλαδή συζητήσεις οι οποίες παραβαίνουν τον κανονισμό και την αντικειμενικότητα αυτής της Επιτροπής. Ένα μέλος το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος μίας επιτροπής θα πρέπει να διαβουλεύεται καθημερινά με τον πρόεδρο και θα πρέπει να όταν εκφράζεται να εκφράζεται προσωπικά και όχι στο όνομα του Κοινοβουλίου. Και εγώ εκείνο το οποίο είπα στην συνάδελφο Μέρτσι είναι ότι θα πρέπει να εκφράζεται προσωπικά. Η κυρία Μέρτσης μου απάντησε ότι όχι, εγώ εκφράζομαι εξ ονόματος όλου του Κοινοβουλίου. Εγώ της είπα ότι δεν μιλάει εκ μέρους του Κοινοβουλίου και αν υπάρχει κάτι κανονιστικό χαίρομαι που τίθεται στις απαραίτητες, στα, στα κατάλληλα όργανα και όχι σε αυτήν την επιτροπή που δεν είναι το κατάλληλο όργανο. Αν υπάρχει λάθος εφαρμογή του κανονισμού από την, από την Προεδρία. Σας παρακαλώ να μου το πείτε γραπτός, δηλαδή να μου το πει γραπτός, συγγνώμη, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω πραγματικά να επιβαρύνω τους παρόντες πολίτες. Συνάδελφε Χάουκεν, εμείς επιβαρύνουμε εδώ τους πολίτες. Είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να εξετάσουμε τώρα. Απαντώ στον συνάδελφο Μακ Μίλαν για το θέμα που έθεσε. Λέω ότι η αναφορά δεν έχει κλείσει. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι στο σημείο 20 διερευνητική επίσκεψη στο Μελάουντα Μούλσε στην Αυστρία και δίνω το λόγο στο συνάδελφο Βίλαντ äh, Ευχαριστώ Πρόεδρε Επιτρέψτε μου Θες να μ' ακούσεις ε, Μακμέλαν επιτρέψτε μου, ε, μια που παρευρίσκεται και ένας άλλος συνάδελφος ε, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Η αναφορά είναι του έτους 2007 και με βάση αυτό το γνώμονα έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Κανονικά το 2008 δεν θα χρειαζόταν ενημερωτικό ε, ταξίδι. Μάλλον δεν μπορέσαμε να το κάνουμε γιατί δεν μας ε, είχαν ενημερώσει αρκετά. Πήγαμε το καλοκαίρι σε μια περιοχή που είναι για χειμερινό σκι. Το 2009 ήταν ε, χρονιά εκλογών και ε, σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι από την Άνοιξη μέχρι το Φθινόπωρο. Εντάξει, είναι χειμερινό σκι ε, εκεί ε, που γίνεται, αλλά υπάρχουν θέματα ζωής και θανάτου. Δεν μπορεί, επειδή έχουμε εκλογέ μια χρονιά το Κοινοβούλιο να παραλύει και η Επιτροπή μα από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο να μην μπορεί να πάει πουθενά ταξίδι. Παρακαλώ πολύ την Πρόεδρο να κάνει κάτι για να ε, αλλάξουν οι κανόνες. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί και η παρέμβαση του Προεδρείου και θα χαιρόμουν να βοηθήσει και ο Αντιπρόεδρος Μακμίλαν Σκότ που συμμετέχει πολύ στην Επιτροπή Μεταφορών και είναι συχνά παρόν. Αυτή ήταν η μία παρατήρηση επί της αρχής. Οι συντονιστές ε, θα πρέπει επιγόντως να ασχοληθούν με το θέμα το, ε, της σύστασης και της σύνθεση των επιτροπών, πώς είναι, πρέπει να είναι παρόντες. Γιατί τελικά ήμουν ο μόνος και μία εξοφίτσιο αυστριακή συνάδελφος, η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα. Όπως και σε κάθε κοινοβούλιο, ε, έχουμε θέματα πιο ευχάριστα και πιο δυσάριστα. Έχουμε και αγκαρίες, τι να κάνουμε. Και πολλοί ενδιαφέρονται να πηγαίνουν στις ωραίες αποστολές και στις προβεβλημένες με πολλά μέσα ενημέρωσης και κάμερες, αλλά υπάρχουν και κάποιες αφανείς και κάπως θα πρέπει να αναγκαστεί η Επιτροπή όταν αποφασίζει να κάνει ε, διερευνητικές ε, αποστολές να πηγαίνουμε και όχι μόνο όταν έρχονται οι κάμερες. Δηλαδή χρειάζεται κάποιο κίνητρο και αν θέλετε το πω και ξεκάθαρα και ένα σύστημα ποινών και κυρώσεων. Ε, δηλαδή πόσοι μπορούν να μεταβούν σε μια τέτοια αποστολή, να υπάρχει ένας μηχανισμός και να εφαρμόζονται αυτά. Τώρα επί της ουσίας. Η έκθεση αυτή είναι προσωρινή. Συμφωνώ όμως με την κυρία Λίχτεμπεργκε. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν κάνει σοβαρά σφάλματα οι τοπικές αρχές. Να θυμίσω περί τίνος πρόκειται. Το όριο των 20 εκταρίων δεν ξέρουμε αν έχει ε, ξεπεραστεί ή όχι για να δούμε αν χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντική ή αν ή δεν χρειάζεται. Στο μεταξύ, εντός παραθέσεως, ε, μείωσε η Αυστρία τα 20 εκτάρια και τα έκανε 10. Δηλαδή, ε, εμείς ελέγχουμε παλιά ε, νομική βάση. Κατά την άποψή μου, τα λάθη που έκαναν οι τοπικές ε, αρχές είναι κάτι που έχει να κάνει με τετραγωνικά και στρέμματα και άρια και όχι εκτάρια δηλαδή. Ε, και ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει ε, να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τις τοπικές αρχές να έχουν διαφορετική προσέγγιση. Εκ των υστέρων σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχετε ξεπεράσει τα 20 εκτάρια. Θα μας στείλουν καταλόγους, λοιπόν, οι τοπικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως χρειάζεται συζήτηση εκτενέστερη και μάλιστα γενικότερα για ε, την οδηγία για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο είναι ακόμα επίκαιρη και πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Επί της ουσίας πρόκειται για το εξή ερώτημα. Η πίστα του σκι συμπεριλαμβάνεται στα εκτάρια, στο εμβαδόν και στην επιφάνεια. Τι λένε οι αυστριακές αρχές και οι δικαστικές αρχές. Στη μελέτη σκοπιμότητας για το περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται μόνο εκείνες οι πίστες του που για να κατασκευαστούν χρειάζεται να αλλάξει το τοπίο και η φύση, η επέμβαση που έχουν άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εγώ που δεν είμαι ειδικό και με, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα τμήμα του οικοπαίδου που χρησιμοποιείται ως πίστα ε, δεν χρησιμοποιείται και πάρα πολύ από την πανίδα. Γιατί είναι ένα ανοιχτός χώρος Αδικημένος από τη φύση, αν θέλετε κιόλας. Και ε, δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει εδώ ε, με τη μελέτη σκοπιμότητας, ε, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και επίσης είναι και το θέμα της επιβάρυνσης. Ε, αν η πίστα χρησιμοποιείται από 50 ανθρώπους την ημέρα, ή 2.000, γιατί διαφέρει και υποδομή εκεί, η υλικοτεχνική, ο αναβατήρας που θα ε, φτιαχτεί και πώς επηρεάζεται και η χλωρίδα και η πανίδα. Και θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί και αυτό το στοιχείο. Ε, στην ουσία πρόκειται για τα εξής δύο θέματα. Και από την Επιτροπή χρειαζόμαστε βοήθεια εδώ. Το θέμα είναι Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για να συμπεριλάβουμε τα μεμονωμένα στοιχεία ενός έργου. Πενταετία για το, για το αν θα έχουν ξεπεραστεί τα 10 ή τα 20 εκτάρια. Για να το πω απλά. Ε, δηλαδή αν είναι αυτό σαλαμοποίηση, πόσο ε, είναι το πάχος της κάθε φέτας του σαλαμιού. Δηλαδή και σε ποιο ε, χρονικό διάστημα εκτείνονται όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη ερώτηση. Σε ποιο βαθμό επιτρέπουμε τα σχέδια αυτά να κατατερματίζονται και να σαλαμοποιούνται και χρονικά αλλά και νομικά. Γιατί είναι διαφορετικές και οι συμβάσεις μετά και τα κομμάτια του έργου. Αλλάζουν και τα νομικά δεδομένα. <laughs> αλλά και τα πραγματικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγάλη ενημέρωση και μεγαλύτερη για αυτό το θέμα και επίσης πώς επιτρέπεται κάτι ε, χρονικά, χωρικά ή νομικά να διονύζεται, να, να πηγαίνει σε μακρους αυτή η διαδικασία. Και επιπλέον, τα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών και ε, σε ό,τι αφορά τις μεσοπρόθεσμες και τις έμες επιπτώσεις. Σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, ας πούμε, δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου νομοθέτη να επιτρέψει να λέει μια χώρα δεν συμπεριλαμβάνω την πίστα ενώ μια άλλη χώρα την περιλαμβάνει και να είναι πιο αυστηρή. Και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά και πολιτική τοποθέτηση. Και θα πρέπει να απαντηθεί και το θέμα ε, τη οδηγία αυτή τη περιβαλλοντική. Μήπω πρέπει να αλλάξει αυτά τα δύο σημεία. Συνοψίζω και πάλι. Δεν πιστεύω ότι οι τοπικέ αρχέ έχουν κάνει σοβαρά σφάλματα και αν, εν πάση περιπτώσει, όχι σε βαθμό που εξάντε να έχουμε καταλήξει ότι ξεπέρασαν τα 20 εκτάρια. Πάντως, η σωστή εφαρμογή τις οδηγία στην Αυστρία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα που θέλω να μου απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά έτσι σε πολύ αδρές γραμμές. Ε, μετά από την ε, επίσκεψη στο Φόραλμπεργκ. Grazie collega Wieland. Ευχαριστώ συνάδελφε Βίλεν, Ο... Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, η κυρία Μαριάν Μιούλεχ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απαντήσω στα τρία ερωτήματα. Θα έπρεπε να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η σχετική οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν ε, τα κριτήρια εκείνα βάσει των οποίων μπορεί να εξλογηθεί ένα σχέδιο να κριθεί μάλλον αν ένα σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή όχι. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε για την αφορά αυτή που πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αυστριακή νομοθεσία περιλάμβανε μια διάταξη που έλεγε που στο μοναδικό κριτήριο το οποίο ίσχυε εκείνη την εποχή στην Αυστρία, δηλαδή ότι μόνο το μέγεθος, η έκταση μιας περιοχής μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο για εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και καταλαβαίνετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ένα πρόβλημα με αυτό, γιατί η οδηγία λέει ξεκάθαρα ότι τα κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται και να εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων το μέγεθος του σχεδίου, αλλά επίσης και άλλα κριτήρια, όπως ε, η φύση της τοποθεσίας ε, κτλ. Ανέλαβε δράση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκίνησε συζητήσεις με τις Αυστριακές Αρχές. Κατά τη διάρκεια των συστήσεων αυτών, η Αυστριακή νομοθεσία τροποποιήθηκε με αποτέλεσμα να μην την υπόψη μόνο το, σχέδιο, το, το μέγεθος του σχεδίου ως βασικό κριτήριο, για το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική δηλαδή μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά άρχισαν να συμπεριλαμβάνονται και άλλα κριτήρια. Επομένω, ένα νομικό πρόβλημα επιλύθηκε. Τώρα να φερθούμε πιο συγκεκριμένα στα γεγονότα. Μετά την τροποποίηση της αυστριακής νομοθεσίας, την ίδια περίπου περίοδο, ο κατασκευαστής αυτού του σχεδίου έκανε διάφορες τροποποιήσεις και αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, μείωσε αρχικά το μέγεθος του σχεδίου και έλαβε επίσης και κάποια άλλα μέτρα που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν τον αντίκτυπο που το σχέδιο αυτό θα έχει στο περιβάλλον. Οι αυστριακές λοιπόν αρχές έκαναν πάλι μια αξιολόγηση για το αν θα έπρεπε δηλαδή να γίνει μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα κριτήρια που λήφθησαν υπόψη δεν ήταν μόνο το σχέδιο του σχεδί, το μέγεθος του σχεδίου, το οποίο είχε άλλωστε μειωθεί, αλλά λάβαν υπόψη τους και άλλα κριτήρια για το αν δηλαδή ε, η νέα αυτή κατασκευή θα δημιουργούσε περισσότερα απορρίμματα, για το αν θα οδηγούσε σε χορύπανση κτλ. Οι αυστριακές αρχές στη συνέχεια λοιπόν κάνανε μια νέα αξιολόγηση και βάσει των κριτηρίων που είχαν επιλέξει και καθότι δεν χρειαζόταν λοιπόν μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφόσον ε, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον δεν ήταν σημαντικός, δεν προχώρησαν λοιπόν στην ε, εκτίμηση αυτή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γίναν όμως οι αλλαγές, όπως σας είπα, στην αυστριακή νομοθεσία. Επανέρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Πώς κάνουμε τους υπολογισμού και τι χρονική περίοδος πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να καθορίσουμε τον αριθμό των εκταρίων που επηρεάζονται. Η οδηγία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω συγκεκριμένο αριθμό ετών Καταλαβαίνετε όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μια λογική εφαρμογή και ερμηνεία τη κοινοτική νομοθεσία. Δηλαδή, η εκτίμηση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη προς την περιβαλλοντική επίπτωση και θα μπορεί γενικά και αόριστα να φέρεται στην αριθμό ετών. Να απαντήσω τώρα στη δεύτερη ερώτησή σας. Αν τα κράτη-μέλη μπορούν να διασπάσουν, αν θέλετε, κάποια μεγάλα project σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επομένως, ένα μεγάλο σχέδιο να παρουσιάζεται ως πολλά μικρά και κατά αυτόν τον τρόπο το μικρό σχέδιο δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για το ζήτημα αυτό, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι δεν επιτρέπεται προφανώς κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα μεγάλο συνεκτικό κατασκευαστικό σχέδιο να κατατέμνεται σε μικρότερα επιμέρους σχέδια μόνο και μόνο για να αποφευχθεί η υπαγωγή στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Βέβαια, η αξιολόγηση πάντα γίνεται κατά περίπτωση, έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σχέδιο που εξετάζουμε κάθε φορά. Πάντως, συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει βάσει των, πληροφοριών που είχε στο συμπέρασμα ότι το μεγάλο αυτό σχέδιο είχε διαιρεθεί σε πολλά επιμέρους μικρότερα σχέδια. Να απαντήσω έτσι και στην τρίτη ερώτησή σας όσον αφορά την κατάτμιση αυτή τη χρονική μεγάλων κατασκευαστικών σχεδίων. Η κατάτμιση αυτή των μεγάλων κατασκευαστικών έργων προφανώς δεν συνάδει με την οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος. Βάσει πάντως των πληροφοριών που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να καταλήξουμε συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο κάνανε εδώ οι αυστριακές αρχές. Μετά τις τροποποίησεις μάλιστα που γίνανε στην Αυστριακή νομοθεσία και μετά τις τροποποίησεις το ίδιο το έργο και μετά τα επιπλέον επίσης μέτρα τα οποία θα ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί η επίπτωση στο περιβάλλον, αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα δεκαετές έργο κατά τη διάρκεια του οποίου θα ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Βάσει λοιπόν αυτών των δεδομένων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ε, οι αυστριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο σφάλμα, ότι κάνανε μη σωστή εφαρμογή ερμηνεία της ε, οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλαντ. Ε, vielen Dank. Also ich Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε αναπερίπτωση έλεγχο βεβαίω. Ο χωρισμός και αυτό το προβλέπουν οι αυστριακοί νόμοι και παραθέτω σε χιονοδρομικά κέντρα οι διατάξεις εφαρμόζονται με το εξής γνώμονα το άθροισμα των δυνατοτήτων που εγκρίθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια συμπεριλαμβανομένων και των ε, διευρύνσεων πρέπει να συμπεριληφθεί. Δηλαδή η πενταετία εκ των υστέρων μου φαίνεται εντάξει. Εξπόστο όμω. Αν το βλέπω όμω εκ των προτέρων και κάνω σχεδιασμό για το μέλλον, ρωτώ πάντα, είναι ένα συνολικό έργο αυτό. Οπότε η πενταετία δεν ξέρω αν άλλε χώρε έχουν μεγαλύτερα διαστήματα. Να σα πω ότι υπάρχει και άλλη αναφορά που αφορά ε, μια γερμανική περίπτωση. Ε, κάτι ε, εγκαταστάσεις για βιοκαύσιμα, για βιοντίζελ. Το σπάσαν το έργο στα δύο για να μείνει κάτω του ορίου. <laughs> Πρέπει να σας πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη δημιουργικότητα και η φαντασία. Και ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή να ε, κάνει μια απογραφή να δει ε, αν αυτό το φαινόμενο είναι περιορισμένο ή μαζικό. Και κάτι άλλο που ρώτησα εγώ και δεν απάντησε καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμή. Τι γίνεται με την πίστα, την ίδια τη χιονοδρομική. Ε, συμπεριλαμβάνεται σε, αυτή, σε αυτό τον υπολογισμό για τα 10 ή τα 20 εκτάρια. Γιατί ε, ο φυσικός νόμος τι λέγει. τα χιονοδρομικά κέντρα που κατασκευάζουν μια στιγμή, λάθος που κατασκευάζουν αναβατήρες ε, διαφόρων τύπων ή ε, ε, η νέα χάραξη πίστας σε χιονοδρομικό κέντρο εφόσον συνδέεται αλλαγή του οικοπαίδου Δηλαδή, όταν φτιάχνουν νέε πίστε που δεν, δεν αλλάζουν τίποτα στο οικόπεδο, δεν αλλάζουν τίποτα ε, στο ε, ε έδαφο, απλώ προσθέτουν τεχνητό χιόνι, α πούμε, δεν αλλάζουν, δεν σκάβουν. Θα έλεγα λοιπόν εγώ ότι δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται αυτές. Αλλά αν έχουμε ένα 20% από τα 100 εκτάρια 20 Βεβαίω επηρεάζεται η φύση και από τους σκιέρ και από τους πάντες. Εφόσον υπάρχει μια ισοπαίδωση της πίστας. Και διερωτώ με αν έχει γίνει σωστά η ε, εφαρμογή της οδηγίας για τις μελέτες ε, περιβαλλον γιατί εξαιρούνται οι χειροδρομικέ πίστες. Και θα ήθελα να μάθω τι κάνει η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία σε αυτό το θέμα, αν έχει ξεπεραστεί ή όχι το ε, όριο. Και εφόσον γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες, τότε θα απαντήσουμε και στο ερώτημα πρέπει να δράσουμε και να ζητήσουμε ε, από ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος κάτι. και θα τους ε, το κάνουμε πάσα αυτό το καυτό θέμα. Ευχαριστώ συνάδελφε Βίλαν για τη δουλειά σας, για την αποστολή που ε, κάνατε και όλα τα προβλήματα, παρά όλα τα προβλήματα που συσσωρεύθηκαν. Κανένας δεν θέλει το λόγο. Περιμένουμε λοιπόν τη γραπτή έκθεση στην οποία θα διευκρινίσουμε τα σημεία τα οποία αναφέρατε και αν θα βαθύνουμε και στο διάλογο με την Επιτροπή. Συγγνώμη, για το τελευταίο θα παρακαλούσα. Ε, και συμφωνεί και η κυρία Λίχτουμπέργκερ. Θα παρακολούσαμε σε αυτό το τελευταίο μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ εξηγευμένη, δεν θέλω σήμερα καν. Αλλά όταν θα έχουμε την τελική έκθεση, παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει προετοιμασμένη και διαβασμένη. Ε, ε, και εγώ αυτό έλεγα. Ε, Εμεί ε, θα συζητήσουμε στο γραπτό κείμενο και τις απαντήσεις που θα μας δώσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Σημείο 19. Κύριε Μπουστινάρου, μπορείτε να το... Αφήστε το σημείο σας για μετά διότι η κυρία Έγκης είπε ότι θέλει να φύγει και μετά να σας δώσω το λόγο. Κυρία Έγκης λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πριν από τρεις εβδομάδες παρουσίασα μια γνωμοδότηση με κάθε λεπτομέρεια. Δεν θα ήθελα λοιπόν τώρα να την επαναλάβω. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι έχετε το σχέδιο γνωμοδότησης μπροστά σας. Θα ήθελα απλώ να πω κάποια πράγματα για τα σημεία τα οποία θίξαμε την προηγούμενη φορά. Ακούσαμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κύριο Διαμαντούρο. Ήταν εδώ επισκέπτη και μα είπε ποια είναι η άποψη για την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την επέκρινε και είπε ότι σε ορισμένα σημεία αποτελεί οπισθοδρόμηση σε σχέση με τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τη χρηστή διακυβέρνηση. Παράλληλα, έκανε μια επικοδομητική καθοδήγηση για το πώ θα μπορούμε να βγαίναμε από το έξοδο το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στον να αποκριθεί στο αίτημά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις καθυστερήσεις αυτές και είπε ότι θα πρέπει να επεξεργαστεί πάρα πολλά στοιχεία προτού απαντήσει η παράδοση της χρυσή διακυβέρνηση και της διαφάνειας θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του νέου κανονισμού, στον πυρήνα του νέου κανονισμού και πρέπει εμείς να υπερασπίσουμε την ε, ακαιρεότητα και την προστασία της ε, ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους κανονισμούς 45 και 1049 και βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρο ότι τα προσωπικά δεδομένα θα μεταφέρονται μόνο στους ε, αποδέκτες εκείνους οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στα απαραίτητα κριτήρια. Ουσιαστικά θα πρέπει να δίνουν την απαραίτητη δικαιολόγηση ή επιχειρηματολογία αν προτιμάτε, η οποία θα καταδεικνύει ότι όντως πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα θεσμικά όργανα θα μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση σε ένα έγγραφο αν η κοινοποίηση του εγγράφου αυτού θέσει κινδύνο την ιδιωτική ζωή ή την, τα εμπιστευτικά δεδομένα ενός ανθρώπου, ενός πολίτη. Θα πρέπει επίσης να εξακριβωθεί αν τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα δικαιολογούν σε κάθε περίπτωση την κοινοποίηση ενός εμπιστευτικού εγγράφου. Είναι σημαντικό οι νέε αυτές πρακτικές να αποτελούν τμήμα της νέας νομοθεσίας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Ακούσαμε τον διαμεσολαβητή, ακούσαμε επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλα τα συμβαλώμενα μέρη αλλά και εγώ ίδια συμφωνώ για το ακόλουθο. Πρώτον, πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τον κανονισμό πρόσβασης στα έγγραφα και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς, ένας κώδικας δεοντολογίας που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της νομοθεσίας αυτής. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα αυτά διάφορες δυνατότητες όπως για παράδειγμα ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή μια συγκεκριμένη συνεδρίαση θα υπάγεται στον κανονισμό αυτό και ότι θα δικαιολογείται ε, η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, η μερική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα καθώς επίσης και η δυνατότητα να υπάρχει μια μη εμπιστευτική περίληψη για κάθε έγγραφο θα είναι κάτι που θα μπορούσε να εξεταστεί. Τον να υπάρχει μερική πρόσβαση σε έγγραφα είναι κάτι το οποίο κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως λέω λοιπόν ξεκάθαρα στην γνωμοδότησή μου, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον ορισμό που δίνουμε στα έγγραφα, γιατί αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κανονισμού. Νομίζω ότι θα, η ιδέα για μια κοινή ομάδα κριτηρίων όσον αφορά την ε, διάθεση ορισμένων εγγράφων, την κατάργηση του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα, θα πρέπει όντως να υπάρχουν τα κριτήρια αυτά, αλλά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλου νομοθετικού εγγράφου, άλλου κανονισμού. Δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να διευρύνουμε τα όρια τα οποία θέτουν οι κανονισμοί. Ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας φιλικός προς το χρήστη κεντρικός κατάλογος εγγράφων, ένα κεντρικό μητρό. Επί της αρχής θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η ιδέα αυτή, στην πράξη όμως απαιτεί τη συνεργασία άλλων των θεσμικών οργάνων για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του συστήματος. Δεν νομίζω επίσης ότι στον κοινοτικό προπολογισμό υπάρχει χρηματοδότηση, προβλέπεται χρηματοδότηση για κάτι τέτοιο. Προτείνω επίσης την ε, γνωμοδότηση να γίνει μια κοινή ε, διεπαφή η οποία θα είναι ε, οικονομικά αποτελεσματική και θα μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις υφιστάμενες τοσελίδες. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ανταλλαγή αυτή απόψεων με τρόπο επικοδομητικό, ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στο ζήτημα αυτό καθ' αυτό και όχι στην όλη προπαγάνδα που το περιβάλλει. Το ΕΛΚ προασπίζει την πρόσβαση στα έγγραφα με τρόπο όμως που δεν θα υπονομεύει την ασφάλεια των πολιτών και ότι δεν θα πρέπει να ακολουθηθούν προπαγανδιστικές, μη ελεγχόμενες πρακτικές. Κατά αυτόν τον τρόπο συνοψίζω την τοποθέτηση του ΕΛΚ και ουσιαστικά αυτόν τον τρόπο συνοψίζω και την δική μου τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Eh, ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσία σας. Την παρουσίασή σας, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καλύπτονται από την προστασία αυτή τα λόμπι, οι ομάδες λόμπι, γιατί ορισμένες προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Νομίζω αντίθετα ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια προς την εργασία τους, να γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι είναι δηλαδή αυτοί που συμμετέχουν στις ομάδες άσκησης πίεσης, στις ομάδες λόμπι. Πολλές φορές έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την ρήτρα privacy της ιδιωτική ζωής για να μην αποκαλυφθούν. Επομένω, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι του μόνου που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι οι πολίτε. Άλλο κανεί θέλει το λόγο. Εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήδη έγινε ανταλλαγή απόψεων στην προηγούμενη συνεδρίαση, επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση τη. Εν γέννη, συμφωνούμε με τι προτάσει που γίνονται από την κυρία Χάνκη στη γνωμοδότησή τη όσον αφορά την παρατήρηση της κυρίας Άουκεν για την ιδιωτική ζωή. Μα η ιδιωτική ζωή δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα. Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων πάντα ζυγίζεται σε σχέση με τα συμφέροντα της διαφάνειας. Αυτό το οποίο λέει ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Λάγκεν είναι ότι η το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ισότιμα δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από τη συνθήκη και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο είπε ότι ο αποχαρακτηρισμός των ε, εγγράφων περιέχουν προσωπικά ε, δεδομένα θα πρέπει να υπάγεται και στους δύο κανονισμούς και όχι μόνο στον έναν κανονισμό. Τον πρώτο δηλαδή για τα προσωπικά δεδομένα. Επομένως τα όσα γίνονται στην πράξη συνάδουν με την απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης είμαι στη διαθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση που ενδεχομένω να έχετε. Ε, μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω μόνο. Υποθέτω και από τις επαφές που έχω εγώ αυτά ακούω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποθέτω λέω ότι ε, βεβαίως η αρχή είναι προς όλους ίση, αλλά δεν είναι ίση ε, οι πολίτες με τα λόμπι. Εμείς θα πρέπει να προστατεύουμε τους πολίτες και βεβαίω για την πρόσβαση στα έγγραφα του κοινού. Εμείς, αν μη τι άλλο, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Αν έχουν την ίδια μεταχείριση τα λόμπε με τους ε, κανονικούς συνήθεις πολίτες, δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. Εξ όσων θυμόμαι εγώ ήταν ασαφής η διατύπωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίζουμε τις διαφορές, όχι μόνο τις αρχές ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στην αρχή. Εδώ όμως οι δύο πλευρές δεν είναι καθόλου ίσες. Βίλαντ. Ο κύριος Βίλαντ. Ωραίο είναι αυτό το σημείο. Ε, για να αποφαθεί κανείς όταν ρωτάει η κυρία Οκεν. Υπάρχουν ε, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ξέρετε, στη ζωή. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε κάποιες αρχές που να μπορούν να εφαρμόζονται. Και όχι αυτός που έχει τα στοιχεία να λέει ότι έχω καλά και κακά στοιχεία και μερικά πρέπει να τα κρύψω ή θέλω να τα κρύψω. Εντάξει, μεγάλη διαφάνεια. Και τώρα αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχουν καλοί και κακοί και από την πλευρά της ζήτησης. Δεν είναι μόνο τα λόμπι, ε, και κάθε μη κυβερνητική οργάνωση τότε λόμπι είναι. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτές συμφέροντα προωθούν. Έτσι δεν είναι. Και αυτό μπορούμε να το δούμε έτσι. Και το άλλο που μπορούμε να δούμε είναι να πούμε ο λόμπις τι κάνει όταν είναι ιδιώτης και το μέλος μιας μη κυβερνητική οργάνωσης και είναι ιδιώτης και πάει σπίτι του και θέλει να έχει πρόσβαση ως ιδιώτης, ως φυσικό πρόσωπο. Θα πρέπει να φυλαχθούμε εκεί. Δεν θα πρέπει ε, να κάνουμε διάκριση μεταξύ καλών και κακών η πλευρά της ζήτησης. Αν μην τώρα μιλήσουμε για ε, θεμητά συμφέροντα και δικαιολογημένα. Αλλιώς θα καταλήξουμε κάπου που ε, θα είναι πιο σκούρα και αδιαφανή τα πράγματα από ό,τι ισχύει μέχρι τώρα. Η κυρία Άουκενμα είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά της Επιτροπής μας το τι θα κάνουμε εδώ στη διαφάνεια. Βεβαίως, όλοι μπορεί να είναι ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα. Και όταν είσαι μίκιο, είσαι Μίκιο. Ε, το ξέρουμε. Ούτε και αυτοί να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Αλλά όταν κάποιος δρά ως λόμπιστ, δεν ε, είναι στην ίδια μοίρα με το μέσο πολίτη. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Και όποιο κάνει δουλειά λόμπι και ασκεί πίεση, είτε είναι η Greenpeace είτε είναι η Bayer, η φαρμακευτική εταιρεία, όλοι πρέπει να είναι διαφανείς. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει να κάνει μόνο με τα φυσικά πρόσωπα, όχι με τα νομικά πρόσωπα. Αυτό το λέει ο κανονισμός 45 του 2001 αναφέρομαστε μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Επομένως, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι επιχειρήσεις δεν καλύπτονται μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της αναθεώρησε αυτού του κανονισμού, προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και είπε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα εφαρμόζεται στα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν δημόσιο ρόλο. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι σε περίπτωση που ένα άτομο το οποίο εκπροσωπεί έναν οργανισμό ή έχει ένα δημόσιο ρόλο, ένα επαγγελματικό ρόλο, τότε δεν προστατεύεται από τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, εκτός και αν υπάρχουν οι συγκεκριμένες εκείνε συνθήκε, εκείνες συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες η αποκάλυψη ταυτότητάς του θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στον ίδιο. Μπορεί να ισχύσει λοιπόν μόνο αν η αποκάλυψη του ρόλου του ή του, ε, του προσώπου του μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για αυτόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάτι τέτοιο γιατί προσπάθησε να ισορροπήσει το δικαίωμα της ε, διαφάνειας με το δικαίωμα προστασίας που έχουν οι πολίτες. Αυτά τα δύο προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε στην αναθεώρηση πρότασης. Κύριε να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, επί της αρχής ή από ιδεολογικής τουλάχιστον πλευράς μπορώ να καταλάβω αυτά τα οποία λέει η κυρία Όκεν. Στην πράξη όμως κάπως φοβάμαι την πρότασή της. Δεν ξέρω πώς μπορούμε πραγματικά να καθορίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο φυσικό πρόσωπο ή το θεσμικό όργανο το πρόβλημα αυτό νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε με τρόπο ξεκάθαρο τη διαφορά ανάμεσα στους μεν και στους δε και στα δικαιώματα μπορούν να έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στα δικαιώματα των φυσικών ατόμων ή και ακόμα και των θεσμικών οργάνων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να οριοθετήσει κανείς ξεκάθαρα τα δικαιώματα αυτά. Και να πω και κάτι ακόμα. Η προθεσμία για την καταβολή τροπολογιών, αν κατάλαβα καλά, ήρθα και σε επαφή με τη γραμματεία. Η προθεσμία λοιπόν είναι η 10η Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Εφόσον λοιπόν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίε στην γνωμοδότηση, έχετε μία εβδομάδα μπροστά σας περίπου για να το πράξετε. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο που θα το συζητήσουμε και στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Παρουσία του κυρίου Χόστινγκς, ο οποίος είναι υπεύθυνο ε, για το Γραφείο Προστασίας των Δεδομένων. Θα το ξαναδούμε λοιπόν το θέμα. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Έγκης. Το λόγο έχει ο κύριος Μπουστινάρου ο οποίος ε, μου ζήτησε να τοποθετηθεί για ένα προηγούμενο θέμα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω να κάνω πάρα πολλές ε, παρατηρήσεις για την ε, πολεμική αυτή που είχαμε την παράθεση στην αρχή της συνεδρίασης. Όσον αφορά την δήλωση της κυρίας Μέρκης, αναφέρεται σε δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην έκθεσή της, στην έκθεση της αντιπροσωπείας η οποία ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σχεδόν με μία αποχή. Δεύτερον, λυπάμαι που λέει χρησιμοποιήθηκε όρος εγκαστρίμηθος στη δήλωση της κυρίας Ματσόνης, η δήλωση της ε, Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών. Νομίζω ότι στο μέλλον όλοι μας θα πρέπει να αποφεύγουμε εκφράσεις οι οποίες ε, λένε πολύ περισσότερα από ό,τι πραγματικότητα έχει συμβεί. Τρίτον, το περιεχόμενο της δήλωσης του Επιτρόπου Μποτόσνικ συνάδει με το περιεχόμενο της δικής μας της έκθεσης, τίποτα το νέο λοιπόν. Και εν τέλει, θα έλεγα ότι η στάση μου σήμερα το πρωί να συνταχθώ ουσιαστικά με το ΕΛΚ και με άλλους για να επιληφθεί το πρόβλημα και να μην επιδεινωθεί ουσιαστικά. Η στάση μου λοιπόν αυτή η θετική είναι ειλικρινής και δεν είχε ως στόχο ούτε να προσβάλλει ούτε να υπονομεύσει την αξία και την εργασία των συναδέλφων μου από τη δική μου ή από άλλες ομάδες. Συνήθως είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τα προβλήματα της χώρας μου. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα ήμουν εξίσου αυστηρός με άλλες χώρες. Γιατί είναι καλό να προστατεύσουμε και λίγο την, να σεβαστούμε μάλλον την ευαισθησία των άλλων και να μην θέτουμε ως στόχο καμία χώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την υπομονή σας και ζητώ συγγνώμη που ξαναπαίρνω τώρα το λόγο. Ήθελα απλώς να αποσαφηνίσω τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι ελπίζω τουλάχιστον θα τελειώσει εδώ η συζήτηση και θα καταφέρουμε όλοι μαζί από κοινού να βρούμε μια λύση, θα καταφέρουμε όλοι να επιλύσουμε το πρόβλημα στην Επιτροπή μας και σε συνεργασία βέβαια με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Εγώ δεν ήθελα να ξαναθίξουμε αυτό το σημείο, αλλά μια που το αρχίζετε να απαντήσω στις παρατηρήσεις σας. Η, την έκθεση δεν την αμφισβητεί κανείς. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει την αποστολή στην καμπανία δεν είναι σωστή η πληροφορία ότι εγώ υπέγραψα το κείμενο, διότι το κείμενο αυτό δεν έχει περάσει ομόφωνα. Τώρα για την απόφαση, την ηλυμένη απόφαση, να σας στείλω τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, ε, που συζητήθηκε το θέμα του να κατέβουμε στην Ολομέλεια με αυτό το θέμα και θα δείτε και από, α, καταγράφω, κάνοντας και απομαγνητοφώνηση δηλαδή τη συνεδρίαση θα διαπιστώσετε ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή απόφαση σήμερα. Να στείλουμε δηλαδή στην έμβη το θέμα, έχουμε μαγνητοφωνημένη τη συνεδρίαση. Μπορεί να είναι λανθασμένη η έκφραση εγκαστρίμηθος. Αλλά κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Διότι κάθε δέκα λεπτά γινόταν μία δήλωση και μετά ξαναδινόταν αυτή η δήλωση από τη συνάδελφο Μέρκης διαφορετικά. Πρόκειται για δηλώσεις όπου η συνάδελφος μιλάει για να αναξιόπιστη κυβέρνηση. Δηλώνει ότι πρέπει να το ξεχάσουν να τα ξεχάσουν τα 145 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τον Μπερλουσκόνη αναξιόπιστο. Αυτή είναι η θέση της αντιπροσωπείας που πήγε στην Καμπανία. Τρεις φορές το είπα. Η συνάδελφος Μέρκης μιλάει εξ ονόματος της ομάδας της και εκφράζει μια πολιτική θέση. Δεν εκφράζει όμως ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε την Εκτελεστική Επιτροπή. Εμείς είμαστε Επιτροπή Αναφορών. Μου φαίνεται λοιπόν σωστό Γι' αυτό λοιπόν εγώ στα Ιταλικά είπα εγκαστρίμηθος που σημαίνει ότι μιλάει για λογαριασμό άλλων. Τους εκπροσώπους δηλαδή του κόμματος της. Αυτή είναι η έννοια του εγκαστρίμηθου στα Ιταλικά. Και όταν κάποιος αναθέτει σε τρίτους να εκπροσωπεί τη χώρα του ε, δεν εκπροσωπεί την Επιτροπή και στη χώρα του. Και η Κόκομπου πάει στην Καμπανία με την προεδρία του κυρίου Ντεματζίστρης. Ενώ εγώ είπα ότι δεν θα προεδρεύσω τις αντιπροσωπείες στην Καμπανία γιατί γιατί δεν θέλω να καπελώσω την αντιπροσωπεία. Γιατί προέρχομαι από εκεί. Και αντίστοιχα σε άλλους αποφάσεις για τη Ρουμανία, για την Πολωνία, εμείς δεν έχουμε εδώ το ρόλο του δικαστή. Εμείς εδώ δίνουμε ένα χέρι στους πολίτες. Και αν ήθελα να ασκήσω πολιτική, τότε θα έλεγα βεβαίως να κάνουμε την έκθεση για την καμπανία, η οποία εδώ και δύο μήνες κυβερνιέται από το δικό μου κόμμα, δύο μήνες. Αυτά κύριε Μπουστινάρου είπα στις συναδέλφους οι οποίες μίλησαν προηγουμένως και κατήγγυλαν την αντικειμενικότητα της Προέδρου, Παρακαλώ λοιπόν να τα βάλετε όλα αυτά γραπτός και να τα κρίνει όποιος πρέπει. Και μετά μπορούμε να απαντήσουμε γραπτός ε, σε όσους εισάγεται το αίτημα. Ελπίζω να εξάντλησα το θέμα και να επανέλθω στην ημερήσια διάταξη και ζητώ συγγνώμη από τους ε, ε, πολίτες που είναι παρόντες εδώ και οι οποίοι μας ακούν εδώ και ώρες να συζητάμε για ένα θέμα καθαρά περιθωριακό. Πάμε στο σημείο 22. 1820 του 2009 του Χωσέ Μαρία Καράσκο Κάνο. Και του δίνω το λόγο. <clears throat> Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Λέγομαι Χωσέ Μαρία Καράσκο και ο συνάδελφος μου Μανουέλ Ρομέρο. Εκπροσωπούμε, μ' ακούτε, ναι, ε, μια ε, ένωση, ένα σύλλογο μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ισπανίας. Εκπροσωπούμε 600.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και ε, αυτοαπασχολούμενους που πλήττονται ε, από την έλλειψη πληρωμών ε, ε, στις νοικοδομήσεις, κατασκευές. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες δεν έχουν πρόβλημα, είναι καλυσμένες. Μετά από 180 ημέρες, 240 ημέρες έχουμε υπερημερίες πληρωμές. Δεν μας πληρώνουν. Γι' αυτό καταφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χάρη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Λαϊκό Κόμμα στη χώρα μας ε, ήρθαμε σήμερα εδώ για να καταθέσουμε αυτή την καταγγελία και την αναφορά. Αυτό που επιθυμούμε είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή Αναφορών να κάνει κάτι για μας, για το σύλλογό μας. Έτσι ώστε στο τέλος των έργων και των κατασκευών και των οικοδομών να μας πληρώνουν, διότι δεν μας πληρώνουν και ε, πτωχεύουν οι μικρές επιχειρήσεις. Έρχεται κάποια στιγμή που βάζουν λουκέτο. Γιατί ε, δεν έχουμε δουλειά, χάνουμε τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας, γιατί ε, είχαμε χρηματοδοτήσει εμείς, προκαταβάλαμε τα ποσά στις τράπεζες και δεν μας πληρώνουν. Και οι δήμοι μας χρωστούν χρήματα και μιλάμε για προθεσμίες τριών και τεσσάρων ε, μηνών υπερημερία. Γι' αυτό πρέπει να καταφεύγουμε σε εξωτερική χρηματοδότηση. Πηγαίνουμε στην τράπεζα και ζητάμε χρήματα και βάζουμε εγγύηση τα σπίτια μας, τα ίδια. Ε, όταν λοιπόν ε, περνούν έξι μήνες χωρίς να έχουμε πληρωθεί οχτώ μήνες, ε, ε, χάνουμε τις εγγύησεις μας που ήταν υποθήκη το σπίτι μας παίρνουν και το σπίτι και μένουμε και στο δρόμο. Οπότε βρισκόμαστε σε ε, μειονεκτική θέση απέναντι στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δίνουμε αυτή τη μάχη τώρα. Αρχίσαμε και χάρη στο Λαϊκό Κόμμα αγωνιζόμαστε για να λυθεί αυτό και με τον νόμο και να μην ευνοούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Επειδή είμαστε μικροί, δηλαδή τι, θα είμαστε σε αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί είναι άνηση η κατάσταση με τις μεγάλες εταιρείες. Ευχαριστώ. Grazie. La parola al ehm, responsabile della Commissione, Deira Robiana Alfonso. Η κυρία Deira Robiana Alfonso. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο αναφερόμενος ε, ιδιαίτερα κατήγγειλε τη μη τήρηση της οδηγίας 2000-35 που είναι η μόνη κοινοτική ε, νομοθεσία ενισχύ για την καταπολέμηση των καθυστερημένων ε, πληρωμών και των επισφαλιών στην ισπανική νομιτάξη. Θα ήθελα καταρχάς εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θυμίσω ότι η εν λόγω οδηγία του 2000 κάθετος 35 έχει μεταφερθεί σωστά στην Ισπανική Ένωμη Τάξη από το νόμο 3 κάθετος του 2004. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση των μεγάλων καθυστερήσεων ε, ε, πληρωμών που περιμένουν οι μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο στις οικοδομές και σε άλλους κλάδους οικονομίας. Και ε, αυτό έχει να κάνει ε, ε, με τους οφειλέτες, μπορεί να είναι και το δημόσιο ή άλλες εταιρείε. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι η σημερινή οδηγία δεν εναρμονίζει την περίοδο πληρωμών, εξού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες εν γέννη. Αυτό ήρθε να το επιβεβαιώσει και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην ε, περίπτωση 380 ε, το 2006 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ισπανίας διότι ε, δεν υπήρχε εναρμόνιση και υποχρέωση εναρμόνισης από την οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε επί κατά του ε, βασιλείου της Ισπανίας γιατί θεωρούσε ότι ήταν υπερβολικά μακρές οι προθεσμίες που έδινε ο νόμος του 2004. Ε, Αλλά επανέλαβε το δικαστήριο ότι δεν υπήρχε εναρμόνιση, ούτε υποχρέωση εναρμόνισης. Όπως ε, παρουσίασε και ο αναφέρομενος, δεν πληρώνονται, δεν καταβάλλονται τόκοι περιμερίας Μα η οδηγία δεν υποχρεώνει τον πιστότη να ε, απαιτήσει τόκους υπερημερίας, αλλά έχει τη δυνατότητα. Όταν έχουμε λοιπόν ε, καθυστέρηση πληρωμών, μπορεί να ζητήσει, ε, αλλά δεν υποχρεούται, επαναλαμβάνω, ο πιστωτής. Κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά την παρακράτηση κυριότητας, στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2035, που μεταφέρθηκε στο νόμο 3 2004 και στο άρθρο 10, ορίζει ότι Ε, Βεβαίω ε, υπάρχει παρακράτηση κυριότητα των αγαθών ε, του οφειλέτη, εφόσον αυτό συνάδει με την εθνική νομοθεσία πάντα. Και σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση σε τρίτους της παρακράτησης κυριότητας, ε, στην υπόθεση 300 ε, του 2005 που είχε προσφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ιταλίας ε, το δικαστήριο όρισε ότι αυτά τα ζητήματα ισχύουν μόνο στην Ισπανία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αναφερόμενος σε ό,τι αναφέρει στην αναφορά του η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αν θεωρούν σκόπιμο ορίζει οδηγία 6 ότι μπορούν να ε, αποκλείσουν ε, τις διαδικασίες ε, πτώχευσης. Αυτό το κάνει και ο αντίστοιχος νόμος. Και τέλος, το τελευταίο που ρωτάει ο αναφερόμενος ως ε, προς την οδηγία για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτή του 2000 αφορά μόνο ε, την ίσπραξη μη αμφισβητουμένων απαιτήσεων και μόνο σε εθνικό επίπεδο. Μη αμφισβητούμενες απαιτήσει, όχι διεθνείς όμως, όχι υπερεθνικές. Γιατί εκεί είναι άλλος κανονισμός, του 2006, ο 1896. Εσείς θέλετε μείωση ε, των προθεσμιών για την απέτηση, για την ίσπραξη. 90 ημέρες είναι σήμερα και η οδηγία ορίζει ότι μπορούν τα κρατη να υιοθετήσουν ή να διατηρήσουν ε, κάποιες διατάξεις που είναι πιο ε, ευνοϊκές για τον πιστότη. Δεν έλαμψε δια τη αποτελεσματικότητα τη βέβαια η παρούσα οδηγία και το γνωρίζει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή τη ήταν προβληματική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό επηρεάζει αρνητικά όλε τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες. Γι' αυτό το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση τροποποίησης τη οδηγία αυτή, 35 του 2000 για να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι κανόνες ε, ω προ την επισφάλεια και ε, τις καθυστερημένες πληρωμές. Στις 21 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ενέκρινε την πρόταση αυτή και χαιρόμαστε. Γι' αυτό και απομένει η ε, τυπική έγκριση του Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Ε, τα κράτη-μέλη διαθέτουν μία διετία για να μεταφέρουν στην ένομή του τάξη. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω μόνο ότι η Ισπανία πρωτοτύπησε Ιουλίου 2010 ενέκρινε το νέο νόμο 15 του 2010 που προχωρεί πολύ περισσότερο από την παρούσα οδηγία ε, ως προς τις θεσμίες πληρωμών. Όπως θα γνωρίζετε εσείς, ο νέος ισπανικός νόμος ορίζει ότι για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ δημοσίων αρχών και ε, ιδιωτικών επιχειρήσεων υπάρχει εναρμόνιση. Οπότε μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να πληρώνουν οι δημόσιες αρχές. Ενώ μεταξύ ιδιωτών ο Ισπανικός νόμος ορίζει ότι η προθεσμία θα είναι 60 ημέρες ε, ε, χωρίς καμία παράταση. Την 1η ε, Ιουνίου του 2013 θα τεθεί σε ισχύ αυτός ο νόμος και ελπίζουμε να δοθεί μια λύση και να διευκολυνθεί η ρευστότητα της αγοράς. Σας λέγω όμως ότι η οδηγία που εγκρίθηκε τώρα εναρμονίζει μόνο τις περιόδους πληρωμών ε, για τις δημόσιες ε, αρχές, 30 ημέρες. Και αυτό σας λέω ε, ότι η Ισπανία πηγαίνει ακόμα παραπέρα και αφορά και τους ιδιώτες. Αν υπάρχει όμως ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών μπορεί να παραταθεί αυτό χωρίς να είναι αυτό εις του πιστωτού για να προστατευτούν έτσι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ε, ότι μπορεί να κλείσει η αναφορά και αυτό προτείνουμε και ελπίζουμε και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στην ομοθεσία τους τη νέα οδηγία το συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τουργάης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ να αρχίσω με τα τελευταία λόγια της Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε σίγουρα είναι να μην κλείσουμε αυτή την αναφορά. Εσείς ε, λέτε ότι πρέπει να την κλείσουμε. Αλλά δίνεται όμως και δίκιο στους εισηγητές λέγοντας ότι έχουν επιχειρήματα για να δικαιωθούν. Λοιπόν, άρα αν κλείσουμε την αναφορά, είναι ε, ζητώντας μας να κλείσετε την αναφορά, αντιφάσκετε στα ίδια σας τα λόγια. Η κρίση σήμερα έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες στα άκρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανησυχία και εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα των αναφερόντων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε όταν ακούγαμε την Κομισιό να κάνουμε, την εξής να κάνουμε μία ερώτηση. Χαιρόμαστε ότι θα λυθεί το πρόβλημα και ότι η Ισπανία θα προχωρήσει και πιο πέρα ε, στην επίλυση, αλλά στο μεταξύ τι έκανε η Κομισιόν όλο αυτό το διάστημα όταν ήξερε <coughs> ότι δεν επληρούτο η οδηγία εκ μέρους της Ισπανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη κάνει παρατήρηση στην Ισπανική κυβέρνηση διαπιστώνοντας ότι δεν εφαρμοζόταν η οδηγία. Σήμερα λέτε ότι θα προχωρήσει και η Ευρώπη και η Ισπανία στην εκπλήρωση κλπ. Και αν λέτε ότι ναι θα εκπληρωθεί θα, εκπληρωθούν, θα τηρηθούν οι όροι της οδηγίας. Οπότε ας μείνει ανοιχτή η αναφορά για να δούμε πώς θα τελειώσει η ιστορία. Και άμα <coughs> τηρηθούν οι όροι της οδηγίας, τόσο το καλύτερο. Θα λυθεί το πρόβλημα των αναφερόντων. Αλλά με το προηγούμενο που έχουμε δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά χωρίς να ξέρουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα δικαιωθούν τα αιτήματα των αναφερόντων και αυτό με το ότι βάσει του γεγονότος ότι τους έδωσε δίκιο η Κομισιόν και ότι η οδηγία δεν ετηρεί στην Ισπανία. Κυρία Γκρουβή. Και εγώ λέω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε, να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και την παρακολούθηση της οδηγίας. Έγιναν ψηφοφορίες τις προάλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι εφαρμογές είναι πάντοτε πολύ δύσκολες. Έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ισπανία. Ο οικονομικός ιστός ε, βρίσκεται στη πλάτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες αυτές και κλείνουν και χάνονται πολλές θέσεις απασχόλησης. Θέλω να τους υποστηρίξω και να παρακολουθήσουμε από κοντά για το πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός στην Ισπανία. Πάντως στην ε, Γαλλία έχουμε μείωση των προθεσμιών πληρωμών, αλλά υπάρχει πάντα πρόβλημα με, τις, ε, με τους θεσμούς. Το δημόσιο πληρώνει πάντοτε αργότερα. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν που ισχύει και σε εμά. Yes, uh, ε, ε. Λοιπόν, εγώ πραγματικά είμαι περήφανη που εκπροσωπώ εδώ τους δύο ετούντες, διότι εκπροσωπούν πολλές οικογένειες, ε, πολύ κόσμο και ένας από αυτούς που είναι εδώ, που βρίσκεται εδώ, πήγε στην Μαδρίτη 600 χιλιόμετρα από το χωριό του, κοντά στο... με τα πόδια και τον είπανε ο Δον Κιχώτη στην Τσικλάνα. Τσικλάνα είναι το χωριό του που είναι κοντά και στο δικό μου χωριό. Λοιπόν, Ήρθε και εδώ στις Βρυξέλλες αυτό που του λέμε δεν κυνηγάει ένα όνειρο, κυνηγάει τα δικαιώματά του. Εμείς ε, λοιπόν θέλουμε να του διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα τα οποία έχει. Ευχαριστώ που η Κομισιόν μας είπε ότι ο νόμος στην Ισπανία θα προχωρήσει. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος Τουργάη δεν, δεν τήρησαν τον νόμο όταν ήταν εκεί που ήταν, πόσο μάλλον άμα πάει και μακρύτερα. Η απελπισία λοιπόν, πρόκειται για απελπισία μικροεπιχειρηματιών που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα και όχι μεγάλες επιχειρήσεις και εκπροσωπούν πολύ κόσμο, όχι μόνο Ισπανούς, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και έχουν την τύχη να είναι παρόντες και να εισακούγονται. Πρέπει να ε, υλοποιηθεί λοιπόν η οδηγία, να εφαρμοστεί, να μεταφερθεί στην Ισπανία να... και να προσαρμοστεί. Πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την αναφορά, να μην την κλείσουμε, διότι γίνονται τέτοιες τρομερές αδικίες που έχουν αφήσει τον κόσμο έρμεο που δεν καταφέρνει καν να πληρώσει τα δίδακτρα του σχολείου των παιδιών του Τι μια άνθρωποι ήτανε. Έχουν καταστραφεί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να είμαστε κουφοί σε αυτού του είδους τα αιτήματα. Και θέλουμε λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ την ε, συνάδελφο. Μου φαίνεται ότι όντως θα μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και το Κοινοβούλιο παρενέβη πριν από μια εβδομάδα για να αναλάβει ακριβώς αυτήν την υπόθεση αλλά θέλουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Παραμένει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη το 23. Πριν δώσω το λόγο στη Στέλλα Βελίκη για την 614 του 2009 Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στεφανή Ρόουτεν που είναι εκπρόσωπος της Βελγικής Προεδρίας. Την ευχαριστώ για την παρουσία της, ευχαριστώ την Βελγική Προεδρία που μας θυμά με την παρουσία της. Η Στέλλα Βελισσή έχει το λόγο. Euh, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας αυτή στην Επιτροπή Αναφορών. Έχω συντάξει μία σύντομη επιστολή στην οποία αναφέρομαι στα βασικά σημεία του ζητήματος. Όπως σας είπα έλαβα κάποιες προτάσεις ε, για να αποσύρω την αναφορά μου ή για να την τροποποιήσω. Η άποψή μου είναι ακόλουθη. Δεν πρόκειται να αποσύρω την αναφορά μου, ούτε πρόκειται να τροποποιήσω. Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα, όσον αφορά τους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού της α, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι αυτοί που ήταν και έχω κάνει πάρα πολλές καταγγελίες και παράπονα και στο Υπουργείο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λαμπυρής. Τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό το οποίο ζητάω είναι ο λογαριασμός φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού να είναι πιο κατανοητός. Να είναι κατανοητός από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πολύ συγκεκριμένες ή επιστημονικές γνώσεις για το ζήτημα αυτό. Ιδίω για το φυσικό αέριο, θα ήθελα να γνωρίζουμε ακριβώς τη μονάδα μέτρησης που καλείται κανεί να πληρώσει. Θα πρέπει να είναι το κυβικό μέτρο και όχι η κιλοβατόρα, η κύβαλα το ημέρα, όπως έχω δει σε κάποιου λογαριασμούς μου στο Βέλγιο. Επίσης θα ήθελα να δοθούν κάποιες λεπτομερείς εξηγήσει στους λογαριασμού αυτούς. Να βλέπουμε δηλαδή σε ένα ξεχωριστό φύλλο τις εξηγήσει που να συνοδεύουν το λογαριασμό Επίσης θα ήθελα και έναν δωρεάν τηλεφωνικό αριθμό όπου θα μπορούν να τηλεφωνούν όλοι οι πελάτες που επιθυμούν να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για το λογαριασμό τους. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς ποιο ποιος είναι ο δρόμος μεταφοράς που καλούμε εγώ να πληρώσω ως πελάτης. Δεν δίδεται καμία πληροφορία προς αυτό. Επίσης θα ήθελα επίσης να γνωρίζω ακριβώς ποια είναι η τιμή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και να γνωρίζω πότε αυξάνεται και πότε μειώνεται η τιμή και γιατί και επίσης θα ήθελα να ε, έχω σε αιτήσια βάση μια δημοσίευση των κερδών της λαμπυρής καθώς επίσης και των άλλων φορέων παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στο Βέλγιο. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ωστόσο η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως στην περιοχή που μένω στο Βέλγιο. Δεν οφείλεται όμως η λαμπυρής για τη βελτίωση αυτή. Είναι η βελγική κυβέρνηση αυτή η οποία επέφερε τις βελτιώσεις. Δηλαδή Στη δικιά μου κοινότητα υπάρχουν πλέον γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει να εξηγήσουν πράγματα όπως ένας λογαριασμός φυσικού αερίου ή ηλεκτρισμού. Και τα γραφεία αυτά μπορούν επίσης να επαληθεύσουν αν έχουν γίνει σωστοί υπολογισμοί στο λογαριασμό. Βλέπετε όμως ότι δεν πρόκειται για πρωτοβουλία της Λαμπυρής, πρόκειται για πρωτοβουλία της βελγικής κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά έχει επιφέρει όντως μία βελτίωση η πρωτοβουλία αυτή και βασίστηκα λίγο στις πληροφορίες που μου έδωσαν τα γραφεία αυτά. Επίσης, θα ήθελα να γνωρίσω καλύτερα πώς έχει ε, η αγορά ενέργειας και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη αγορά φυσικού αερίου. Από όσο γνωρίζω εγώ, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και το φυσικό αέριο τελικά, η τιμή του εξαρτάται πάρα πολύ από την τιμή του πετρελαίου. Για μένα, οι δύο αυτές πηγές ενέργειας είναι εντελώ διαφορετικές. Για ποιο λόγο θα πρέπει το φυσικό αέριο να εξαρτάται από την τιμή του πετρελαίου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει μια ξεχωριστή αγορά φυσικού αερίου. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη είναι η ακόλουθη. αν δεν έχει γίνει η απελευθέρωση της αγοράς όπως θα έπρεπε για το φυσικό αέριο, για ποιο, για ποιο λόγο τουλάχιστον δεν υπάρχει μία μέγιστη τιμή του φυσικού αερίου έτσι ώστε οι διακυμάνσεις να περιορίζονται κάτω από αυτό το ανώτατο πλαφόν. Αυτά είχα να σας πω. Επί της αρχής εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση όσον αφορά τους λογαριασμούς φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος της λαμπύρης. Εξακολουθούν να είναι ακατανόητοι αυτοί οι λογαριασμοί. Ακόμα και όταν α, τηλεφωνώ Ακόμα και όταν τηλεφωνώ στη Λαμπυρή, πάντα τέτοια προβλήματα συναντώ. Δεν μου δίδεται καμία εξήγηση. Η γραμμή εξυπηρέτησης πελατών υποτίθεται ότι ε, είναι εκεί για να μας βοηθήσει και καταλήγω τελικά εγώ να τους λέω τι πληροφορίες χρειαζόμαστε εμείς οι πελάτες. Ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Βελίκη. Απαντήσαμε στη αναφορά αυτή πέρσι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Η αναφερόμενη είχε πει ότι ήταν δύσκολο να ε, απευθυνθεί στην εταιρεία αυτή. Το έκανα ίδια και μου ε, χρειάστηκαν ακριβώς τρία λεπτά. Δεν ήταν αυτόματος τηλεφωνητής, ήταν ε, άνθρωπος που μου απάντησε. Συχνά κατηγορούνται οι εταιρείε ότι δεν έχουν σωστή εξυπηρέτηση πελατών. Εγώ μίλησα με κάποιον μετά από τρία λεπτά, το χρονομέτρησα. Ε, στη μονάδα μου για την εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήλεγξα επαλήθευσα τα όσα μας λέτε γιατί η δουλειά μας είναι να σας απαντάμε επί της ουσίας και μου απάντησαν ότι οφείλατε πάρα πολλά χρήματα στην εταιρεία μη πληρώνοντας τους λογαριασμούς σας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2009 τροποποιήθηκαν οι οδηγίες 2009-72 ε, και 73 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ε, εσείς οι βουλευτές ορίσατε ε, τι θα πρέπει να αναφέρετε κατελάχιστον σε ένα τιμολόγιο παροχής ενέργειας. Αυτό αναφέρεται και στο παράρτημα 1 ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ότι στην εμπορική σχέση μεταξύ πελάτου και εταιρεία υπάρχουν κάποιε ελάχιστε απαιτήσει του κοινοτικού δικαίου που βεβαίως ε, εκπονήθηκαν ε, μετά από στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο γιατί δεν είναι συναπόφαση προφανώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εταιρεία Λαμπύρης, για να επιστρέψουμε, είναι μια μεμονωμένη ιδιωτική περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της εσωτερικής γενικής διεύθυνσης Υγεία και Προστασία των καταναλωτών έχει προβεί σε συστάσει. Το οποίο όμω αυτό δεν είναι νομοθεσία. Η νομοθεσία χαράστε και αποφασίζεται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Εμεί συστάσει κάνουμε στι εταιρείε ενεργειακέ. Οι συστάσει είναι και δημόσιε, εγκρίθηκαν πέρσι από το Φόρουμ του Λονδίνου, που είναι ε, ο αρμόδιο φορέα και έχει συσταθεί προτριετία και ο υπουργό Μανιέτ ε, Βελγικής Προεδρία, μάλιστα μα είναι χάρη στην ε, Εκτελεστική Επιτροπή για τη θέσπιση αυτού του οργάνου και εκεί αν θέλετε εξετάζουμε περισσότερο την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και κάνουμε συστάσεις χωρίς αυτό να έχει δεσμευτική ισχύ, δεν είμαστε δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στο Βέλγιο, η βελγική κυβέρνηση δημιουργήσε και τη θέση του διαμεσολαβητή, του ενεργειακού και σας απάντησα σε αυτό. Είναι ανεξάρτητος φορέας, ανεξάρτητος και από τις εταιρείες προφανώς, αλλιώς δεν θα ήταν αποτελεσματικός και ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του κοινοτικού δικαίου ε, που εγκρίνατε πέρσι. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου, βεβαίως αυτό το θέμα ξεπερνάει κατά πολύ το πεδίο της αναφοράς γιατί έχουμε ένα πρόβλημα τιμολογίου και ενφερόμενοι μας κάνει ερωτήσεις τώρα για το πώς λειτουργεί η αγορά φυσικού αερίου και πώς ε, συνδέεται στο βέλιο Για κάποιον δηλαδή που δεν μπορεί να διαβάσει το λογαριασμό του ρεύματος, αυτό είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και η αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι γνωστή. Δεν υπάρχει η αποσύνδεση αυτή τη στιγμή ε, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τη διαχείριση και ορισμένα τμήματα της αναφοράς για τη λειτουργία της αγοράς αερίου νομίζω ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό ε, τη λειτουργία της εταιρεία Λαμπύρης που ε, παρέχει και φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για να απαντήσω. Ο συνάδελφος Κυρία Πρόεδρε, το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται μόνο στο Βέλγιο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε και αλλού. Θα έλεγα ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Η τιμολόγηση του φυσικού αερίου γίνεται με βάση τις ε, κιλοβατόρες. Αυτή είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας. Δεν πρόκειται για μονάδα μέτρησης όγκου όμως του φυσικού αερίου το οποίο χρησιμοποιείται εκτός και είναι κανείς μηχανικός, εμπειρογνώμονας ή φυσικός, είναι πολύ δύσκολο για τον απλό πολίτη και πελάτη να καταλάβει την πραγματική αξία του χρησιμοποιημένου φυσικού αερίου, γιατί όλα τα μηχανήματα τα οποία καταγράφουν τη χρήση φυσικού αερίου χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο δεν υπάρχει κανένας πίνακας αντιστοίχηση στη συνέχεια, προκειμένου να καταλάβει κανείς σε τι ενέργεια αντιστοιχούν αυτά τα κυβικά μέτρα, ο όγκος δηλαδή που έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης, η μετάφραση έπειτα του αερίου αυτού σε κιλοβατόρες έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου όγκου, ενός συγκεκριμένου όγκου φυσικού αερίου. Πολλές φορές στη χώρα μου, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το χρησιμοποιούμενο φυσικό αέριο και όγκο του φυσικού αερίου συρρυκνώνται και πολλές φορές ε, και η ίδια η ενεργειακή απόδοση, αν θέλετε, αυτού του όγκου φυσικού αερίου μειώνεται. Παρ' όλα αυτά ο πελάτης συνεχίζει και πληρώνει την ίδια αξία, την ίδια ενεργειακή αξία. Οι πελάτε και οι καταναλωτέ δεν το γνωρίζουν αυτό. Μίλησα με πυρογνώμονε, με μηχανικού, οι οποίοι μου είπαν ότι και αυτοί δυσκολεύονται πάρα πολύ όταν πρέπει να περάσουν από του κιλοβατόρε στα κυβικά μέτρα, όταν πρέπει να κάνουν δηλαδή αυτή την αντιστοίχηση. Φανταστείτε λοιπόν πόσο περίπλοκα φαίνονται τα πράγματα για τον απλό πελάτη, ο οποίο λαμβάνει λογαριασμό και δεν μπορεί να καταλάβει τελικά τι διαβάζει. Τα πράγματα όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια ενδεχομένω είναι κάπω πιο απλά. Τα ε, μηχανήματα μέτρηση για το φυσικό αέριο καταγράφουν μόνο, μετράνε μόνο και ειδικά μέτρα. Θεωρώ ότι οι πελάτες στη συνέχεια χρειάζονται μια αποκωδικοποίηση για να καταλάβουν τελικά ποια ήταν η κατανάλωσή τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από όλου του Ευρωπαίου πολίτε να έχουν τι γνώσει επιστημόνων, μηχανικών, φυσικών, χημικών, προκειμένου να καταλάβουν ακριβώ ποια είναι η κατανάλωσή του, ούτε έχουν τα απαραίτητα εργαλεία, τα μηχανήματα που θα του επέτρεπαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητάμε να βοηθήσει τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ νέο μέλος και αναπληρωματικό μάλιστα. Ε, δεν θέλω να σας δυσκολέψω τις εργασίες της Επιτροπής. Εκτιμώ πολύ την, ημερήσια, ε, την πρόεδρο συγγνώμη, που θέλει να, να τηρεί την ημερήσια διάταξη. πρέπει να σας πω ότι είμαι νομικός και δικηγορό και ε, επιθυμώ να μιλήσω για τη συγκεκριμένη αφορά. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση που συμμετέχω στην Επιτροπή εδώ και είναι σαφές ότι τα μέλη είναι νομικοί και μη νομικοί. Πολλές φορές θα ήταν πιο εύκολο να εξτάζουμε τα θέματα αν ξέραμε περισσότερα πράγματα. Στο συγκεκριμένο δεν μας έχουν απαντήσει ε, και κανείς δεν μας είπε γιατί οφείλει η κυρία 4.500 ε, ευρώ στην εταιρεία ε, Λαμπύρης. Διότι δεν πρόκειται εδώ για παράβαση των κοινοτικών κανόνων, παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Io ε, ευχαριστώ. Η απάντηση της Κομισιόν είναι σαφέστατη. η οποία λέει ότι είναι εθνική αρμοδιότητα και ότι υπάρχει εθνικός διαμεσολαβητής όπου να απευθυνθεί η αναφέρουσα. Βέβαια υπάρχει και αυτό το κατανοητό το οποίο, επιχείρημα που μας ανέφερε ο κύριος στην Άρου Σημεριζόμαστε όλοι λοιπόν την θέση της Κομισιόν. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, κλείνει αυτή η αναφορά και παραπέμπω στις εθνικές αρχές την επίλυση του προβλήματος της κυρίας Βελίκη. Πάμε στην επόμενη τώρα, 762 του 2009, της Γιολάντα Σεσβιώτ, και δίνω το λόγο στην αναφέρουσα. Είναι παρούσα. Καλημέρα. Λέγομαι Γιολάντα Στεμπιότ και κατέθεσα μία αναφορά κατά της Ryanair. Πέρυσι αντιμετώπισα προβλήματα με ακύρωση πτήσεων και 45 λεπτά χρειάστηκα σε ένα επιπληρωμή τηλέφωνο ε, για να μου απαντήσουν με ένα ευρώ το λεπτό για να κυρώσω την πτήση επιστροφής και αναρωτιέμαι γιατί χρησιμοποιούν αυτά τα επιπληρωμή νούμερα για τις απλές πληροφορίες και όχι νούμερα με με νορμάλ ε, τιμολόγηση όπως κάνουν οι άλλες, οι άλλες εταιρείες. Πρέπει να σας πω ότι οι όροι ακύρωσης στο, στην ιστοσελίδα της Ryanair δεν είναι πολύ σαφής δεν μας επιτρέπουν να κυρώσουμε ή να έχουμε πληροφορίες πριν από την κράτηση πιστεύω ότι τα δικαιώματά μας των καταναλωτών δεν είναι σεβαστά από αυτήν την εταιρεία και ζητώ να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά ούτως ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μετά την πώληση και των υπηρεσιών της Ryanair για τους μελλοντικούς της επιβάτες. Κομισιόν. Άντζελο Γκρέκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο είναι τα βασικά θέματα. Το κόστος και ε, ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η τεχνική βοήθεια, υποστήριξη. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια φτηνά. Ε, όμως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει να είναι ενήμερος ο πελάτης για το κόστος αυτό. Υπάρχει αυτή η οδηγία, την έχουμε συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποχρώνει την αεροπορική εταιρεία ε, ή την όποια εταιρεία να ενημερώνει ε, τους πελάτες ε, για οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και το κόστος αυτής. Και με ποιον τρόπο παρέχεται και ποιες είναι οι συνθήκες, αυτά θα πρέπει να είναι σαφή όλα κατά τη διάρκεια της κράτησης ή ακόμα και πριν λάβει χώρα η συναλλαγή. Επίσης, έχουμε μια οδηγία που ε, προστατεύει τους καταναλωτές ε, από αθέμητες πρακτικές ε, εις βάρος του καταναλωτού και υπέρ της εταιρείας. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει μόνο αυτή η ακριβή τηλεφωνική γραμμή για παράπονα και καταγγελίες, αυτό μπορεί να προσβληθεί με βάση μια οδηγία για την ενημέρωση των καταναλωτών. Τώρα όμως η εφαρμογή αυτών ε, των ε, οδηγιών και της νομοθεσίας είναι θέμα των κρατών μελών. Έχει μεταφερθεί η οδηγία αυτή στα κράτη-μέλη και υλοποιείται, εφαρμόζεται. Ε, είχαν λοιπόν την ευκαιρία τα κράτη-μέλη να προσφύγουν κατά τέτοιου είδους πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν συστήνει στην αναφερομένη να φέρει το θέμα ε, υπόψη ε, των αρμοδίων εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες σταθμίζοντας ε, την κατάσταση να αποφαθούν αν και κατά πόσο έχουν παραβιαστεί, έχουν γίνει σεβαστοί οι κανόνες για τη σωστή και θεμητή λειτουργία της αγοράς σε αυτό το τομέα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να ζητήσετε ε, σε ε, σημείο ε, ενημέρωσης των Ευρωπαίων καταναλωτών περισσότερες πληροφορίες. Πρόκειται για ένα δίκτυο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθάει τους πολίτες που έχουν τέτοια προβλήματα σε διασυνοριακές συναλλαγές. τύπου κράτησης στο διαδίκτυο. Και επίση υπάρχει ένα κανονισμό για την προστασία των καταναλωτών και συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών, ακριβώ σε περίπτωση διεσυνοριακών προβλημάτων. Και έχει και βελτιωθεί και διευρυνθεί αυτό, γιατί τώρα οι αρχές είναι υποχρεωμένες να ε, συνεργάζονται και οι δικαστικέ αρχέ και οι εθνικέ αρχέ στην Πολωνία, πούμε, θα μπορούσαν να ζητήσουν ε, βοήθεια, η δικαστική συνδρομή ε, από τις Ιρλανδικές. Δεν ξέρω που εδρεύει η ε, Ryanair σε σχέση με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Και να γίνουν απαραίτητες έρευνες για να σταματήσουν τέτοιου είδους πρακτικές. Συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθήστε πρώτα να λύσετε αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο, όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατάλληλα εργαλεία για επίλυση. Θέλει κανείς το λόγο. Η κυρία Γκρινή. Ναι, καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη είναι τα αρμόδια για την επίλυση του προβλήματος. παρόλα αυτά να μείνει ανοιχτή αναφορά. Γιατί η Ryanair είναι μια εταιρεία που προτείνει πολύ χαμηλές τιμές. Όταν όμως βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην πραγματικότητα, καλεί τον πελάτη Ryanair να πληρώνει τα πάντα στη συνέχεια και συνεχώς οι πελάτες συναντούν δυσκολίες και στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγές κατά της Ryanair. Καταλαβαίνω την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι η αναφέρουσα θα μπορέσει να κάνει προσφυγή και στο εθνικό επίπεδο. Εγώ αυτό που θέλω είναι να γνωρίζουμε ουσιαστικά τι πρόκειται να κάνει συνέχεια αναφέρουσα, τι απάντηση θα της δοθεί, τι άλλε δυνατότητε θα έχει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να μιλήσω ως πρώην δικηγόρος. Ε, επί αναφοράς της ίδιας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη ΡΕΝΕΡ αλλά εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα η Ισπανία και η ε, Γαλλία απαγορεύουν τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά ε, υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη όπου δεν υποχρεούνται οι εταιρείε να εξυπηρετούν τους πελάτες τηλεφωνικά με κανονικές τιμές και όχι με αυξημένο τιμολόγιο. Σε επίπεδο κρατών μελών λοιπόν πρέπει πρώτα να λυθεί το ζήτημα και μετά να ε, καταπολεμούνται οι αθέμητες πρακτικές για την προστασία των ε, πελατών. Αυτό είναι εθνική νομοθεσία. Μου φαίνεται να κατάλαβα ότι θα πρέπει η Ενεπέρουσα να κάνει μία αίτηση στις τοπικές αρχές και θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά για να δούμε τι απαντήσεις θα λάβει η αναφέρουσα. Πάμε στο 21 στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, ε, ο συνάδελφος Χέφνερ έχει το λόγο που εκπροσωπεί και την κυρία Γουόλης η οποία χρειάστηκε να φύγει. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω ένα μικρό κρυολόγημα και σας ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου που είναι λίγο βραχνή. Έχουμε τώρα μια μεγάλη ευκαιρία ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών, να τις δώσουμε σάρκα και οστά, δηλαδή να έχουν οι πολίτες πλέον οι πολίτες την ευκαιρία να κάνουν ε, προτάσεις, ιδέες, αλλά να φέρουν και προβλήματα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα θεμέλια τα έχει βάλει η συνθήκη τη Λισαβόνα και αυτό τον καιρό ε, συζητούμε ε, το πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Είναι τέσσερις οι εισηγητές, δύο της ε, συνταγματικής και δύο της Επιτροπής Αναφορών. Ο Αλέ Λαμασούρ, η Ζήτα Γκουρμάη από την Επιτροπή Συνταγματικών και από εμά η κυρία Γουόλης και εγώ με διάφορους και οδησηγητές, με πάρα πολύ καλή συνεργασία μια σειρά συνεδριάσεων έχουμε ήδη δεξαγαγή και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους σκιώδεις ηγητές της Επιτροπής Αναφορών που συμμετέχουν πάντα ενεργά ε, σε αυτή τη συνεδρίαση. Ε, δεν μπορεί παρά να βοηθήσει την υπόθεση. Τώρα, χρονικά, ενημερώνουμε τη συνεδρίαση αυτή για την κατάσταση των συζητήσεων ε, και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών θα καταθέσουμε και έκθεση για να τη συζητήσουμε και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο μπορούμε να καταλήξουμε. Πώς έχει το σχέδιο να προσπαθήσουμε ε, να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή, θα διαπραγματευθούμε επίσημα με το Συμβούλιο και την Επιτροπή μόλις εγκριθεί από τις Επιτροπές η έκθεση για μια κοινή λύση και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια κοινή λύση και τελικά στην Ολομέλεια να περάσει το Δεκέμβριο. Βεβαίω με την επιφύλαξη ότι θα υπάρξει μια τέτοια συνολική κοινή λύση. Προ το παρόν έχουμε πολλέ ανταλλαγέ απόψεων και μας έχετε διαβεβαιώσει κι εσείς συνεχίζουν οι άτυπες επαφές και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ουσία. Θα ήθελα να σας αναφέρω μόνο τα σημαντικότερα ε, της δικής μας έκθεσης, για τη δική μας Επιτροπή ενώ αναφορών. Ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό συμπίπτει με τα όσα εκπονεί η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων με μικρές αποκλήσεις. Εγώ θα επικεντρωθώ όμως στα σημαντικότερα για τη δική μας Επιτροπή Αναφορών. Το σημαντικότερο για μας είναι το θέμα ε, της έγκρισης ε, του παραδεκτού ε, μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε τρία εμπόδια, τρεις φάσεις. Πρώτον, μία υπογραφή Μία υπογραφή, ένας πολίτης ζητάει κάτι και αν ε, είναι σοβαρό, αν δεν είναι καταχρηστικό, αν δεν ε, αντιτίθεται κατά των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά άλλα. Αν όλα αυτά ισχύουν και συντρέχουν, τότε καταχωρείται η πρωτοβουλία αυτή και ακολουθεί η δεύτερη έγκριση. Ε, αυτή τη στιγμή έχει συλλέξει 300.000 υπογραφές, θα πρέπει για μερικούς μήνες να σταματήσει η διαδικασία και μετά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα το ελέγχει αν όλα αυτά είναι παραδεκτά από πλευράς νομικής και μπορούν να συνεχίσουν. Αλλιώς από την αρχή ή να βαγεί η όλη προσπάθεια. Εδώ το Συμβούλιο αντί για 300.000 υπογραφές προτείνει 100.000 υπογραφές. Και μετά η τρίτη επαλήθευση και δεσμευτική είναι εφόσον έχουν συλλεγεί ένα εκατομμύριο υπογραφέ και πάλι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ελέγχει, να δει αν θα το υποστηρίξει, αν θα δώσει συνέχεια, αν θα υπάρχει πολιτική υποστήριξη για νομοθεσία, οδηγία ή κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη με τρία στάδια, τρεις φάσεις, να γίνει λιγότερο γραφειοκρατική, πιο φιλική για τον πολίτη, πιο light με δύο φάσεις μόνο, μία στην αρχή και μία στο τέλος. Και αυτό το μεσαίο στάδιο των 300.000 ή των 100.000 υπογραφών να καταργηθεί. Γιατί δεν έχει νόημα τώρα μεσού τη διαδικασία ξαφνικά να λέμε όπ, σταματήστε λίγο να δούμε, να κοιτάξουμε και μετά μπορείτε να συνεχίσετε. Ε, λοιπόν, και είπαμε όμως στην αρχή όχι μία υπογραφή μόνο, αλλά επτά. Να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι δεν είναι ο κάθε πικραμένος που έρχεται να πει τον πόνο του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στέλνει ένα email επειδή ε, έχει ζητήματα και ξαφνικά αυτό να καταχωρείται ως πρωτοβουλία πολιτών. Όχι. Να είναι 7 και μάλιστα όχι από μια χώρα, αλλά από 7 κράτη-μέλη να έχουν προβληματιστεί, να είναι πραγματική πρωτοβουλία που έχουν σχεδιάσει. Δηλαδή, να φτάσει και σε 100.000 υπογραφές, έτσι. Ε, μετά όντως θέλουμε να ελέγχεται αν κατά πόσο η ε, πρωτοβουλία αυτή ε, είναι επιτρεπτή και παραδεκτή στα πλαίσια των συνθήκων, δεν αντιτίθεται δηλαδή στις βασικές αρχές της Ένωσης, όπως λέει το άρθρο 2 της Συνδίκης Λισαβόνας, και επίσης εάν πρόκειται για ένα αντικείμενο για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας και μπορεί να το ασκήσει. Αν συντρέχουν όλα αυτά, μπορούν να αρχίσουν να μαζεύουν υπογραφές. Και η δεύτερη επαλήθευση και ε, η ε, δεσμευτική είναι εφόσον έχουν συλλεγεί 100.000 ε, υπογραφές. Αυτά όλα τα θεωρούμε πιο πρακτικά, πιο εφαρμόσιμα. Ε, συζητήσαμε με πολλές κυβερνήσεις, πολλές πρωτοβουλίες για την Ευρώπη και θεωρούμε ότι, και είδαμε ότι είναι πολύ μεγάλη υποστήριξη και μας ε, τράβηξε και την προσοχή αυτό, είναι αξιοπρόσεκτο. Ε, γιατί και στις κυβερνήσεις που τελικά θα κληθούν να εφαρμόσουν όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι άλλο τώρα. Ποιος έχει δικαίωμα να ξεκινάει η πρωτοβουλία. Μόνο νομικά, ε, φυσικά συγγνώμη πρόσωπα, όχι νομικά πρόσωπα. Δεν θεωρούμε ότι είναι αυτό εργαλείο για κόμματα, για συλλόγους, για ενώσεις, για επιχειρήσεις για εταιρείε. Είναι για τους πολίτες, για τα φυσικά πρόσωπα. Άλλωστε αυτό το ορίζει σαφώς. Είναι το για πολίτες, citizens, όχι companies και τέτοια πράγματα. Ε, και ε, εμείς επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Μόνο φυσικά πρόσωπα να έχουν το δικαίωμα. Επίσης, οι πρωτοβουλίε αυτές που συλλέγουν υπογραφέ να έχουν και διαφάνεια υποχρεωτικά ως προς τη χρηματοδότησή τους. Δηλαδή, Ποιο του χρηματοδοτεί, ποιο βρίσκεται από πίσω, ποιο το υποστηρίζει και με γενναία ποσά. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο, ε, ένα ποσό, όχι το κάθε γραμματόσημο ή δεν ξέρω κάθε δαπάνη τη τάξεω του ενό ευρώ να δικαιολογείται, αλλά από χίλια ευρώ και πάνω χρειάζονται παραστατικά. Ποιο σα πληρώνει να κάνετε αυτή την πρωτοβουλία. Το τρίτο. ποιο μπορεί να υπογράφει τώρα μια τέτοια ε, πρωτοβουλία πολιτών. Και εδώ εμείς προτείνουμε κάθε Ευρωπαίος και Ευρωπαία από την ηλικία των 16 ετών και μετά. Εδώ διαφέρει λίγο η πρόταση από εκείνη τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει μόνο όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Θα γνωρίζετε όλοι, είμαστε μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι το δικαίωμα του αναφέρεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εδώ ηλικιακός και κατά ε, την εμπειρία μας αυτό δεν οδήγησε σε κανένα πρόβλημα με την ε, πρωτοβουλία των πολιτών λοιπόν εμείς δεν δημιουργούμε κανένα μέσο ή κανένα εργαλείο ε, υποχρεωτικής εφαρμογής, δεν είναι ψηφοφορία. Προτάσει κάνουν οι άνθρωποι, έχουν μια πρωτοβουλία και την προβάλλουν. Ε, γι' αυτό δεν θέλουμε υπερβολικά να περιορίσουμε αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας κάνει καλό και σε εμά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν πιο νέοι ε, πολίτες να έχουν τη δυνατότητα ε, να εκφράζουν τα μελήματά τους. Εξού και το 16. Από πόσα κράτη-μέλη τώρα θα πρέπει να προέρχονται αυτές οι υπογραφές. Είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα και επιθυμία από όλα τα κράτη-μέλη. Στο σχέδιο υπάρχει και άλλο εμπόδιο. Στη συνθήκη εννοώ. Ε, γίνεται λόγος για σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Ε, για αρκετές υπογραφές. Εμείς προτείνουμε ο σημαντικός αριθμός να γίνει ένα πέμπτο των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα τρίτο. Ε, κάπου θα διαπραγματευτούμε στο τέλος. Ε, σημαντική άλλη ερώτηση. Από ποιο χρονικό σημείο και μετά ακυρώνονται οι απογραφές. Στο ε, σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν μια ε, καταληκτική ημερομηνία έτσι αρκετά χονδρική μετά από 12 μήνες λέει. Αλλά σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία για συλλογή υπογραφών διασυνοριακά σε διάφορες γλώσσες και σε διάφορες χώρες και με εθνική δυνατότητα, όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ λίγο το διάστημα 12 μήνες. Αν σε πολλές χώρες, σε πολλές γλώσσες διασυνοριακά και δεν είναι και πάντα online αλλά και offline μπορεί να να μαζεύει υπογραφές έτσι. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε ανθρώπους που δεν ε, κινούνται στο διαδίκτυο από τη συλλογή υπογραφών. Όχι. Οπότε το διάστημα των 12 μηνών μας φαίνεται πάρα πολύ λίγο μικρό και ζητούμε 18 μήνες. Α, παρένθεση. Η Επιτροπή Ελευθεριών του Κοινοβουλίου μας ζήτησε 24 μήνες διετία σε αντίθεση με εμά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 12 μήνες, ένα χρόνο, εμείς 1,5. Ένα άλλο τώρα αποφασιστικό ερώτημα για την πρωτοβουλία των πολιτών, ίσως και το αποφασιστικότερο θα είναι και στο τέλος τι θα γίνει. Όταν συλλεγούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, φανταστείτε τη ζυγαριά ας πούμε, τώρα δημιουργούμε ένα κανονισμό και μια ρύθμιση που, πώς να το πω, δημιουργεί πολλούς κανόνες που θα πρέπει να σέβονται οι πολίτες, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να γίνει αυτή η πρωτοβουλία και τι να τηρούν. Ένα εκατομμύριο υπογραφές σε τουλάχιστον ένα πέμπτο των κρατών μελών, ε, με διάφορους όρους και προϋποθέσεις. Ωραία. Και τώρα οι ε, πολίτες θα ρωτήσουν και το άλλο τάση της ζυγαριάς δηλαδή τι έχει. Εντάξει τα κάναμε όλα εμείς αυτά, εσείς τι κάνετε τις υπογραφές. Θα μας στείλετε γράμμα, θα μας ακούσετε, θα συζητήσετε σοβαρά και θα λάβετε υπόψη αυτά που λέμε. Και από την αρχή είπαμε ότι αν κάποιος καταφέρει να μαζέψει ένα εκατομμύριο υπογραφές, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καλεί τους πολίτες, όχι το ένα εκατομμύριο, εκείνους που ξεκίνησαν, ε, τους εμπνευστές πρωτοβουλίες και σε ε, δημόσια ακρόαση να τους ακούσει και να συντηθούν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Γιατί αυτό είναι το ελάχιστο που τους αξίζει και τους οφείλουμε και θα πρέπει να τους εγγυηθούμε. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος να συμφωνήσει. Είναι στη διακριτική της ευκαιρία και καλά κάνει και είναι. Το λέγανε και οι συνθήκες. Αλλά η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να κάνει ό,τι θέλει. Ε, ε, χρειάζεται μια διαδικασία γιατί η δημοκρατία λειτουργεί μέσω από διαδικασίες και οι πολίτες, ακόμα και εμείς, δεχόμαστε μια αρνητική ε, απόφαση, μια απόρριψη καλύτερα αν μας έχουν ακούσει. Γιατί αν δεν μας έχουν ακούσει καν, σου λέω, γιατί μου το απορρίπτεις αφού ούτε καν άκουσες τι θέλω. Για να μην δημιουργούμε μεγάλες απογοητεύσεις και ε, αποκαρδιώνουμε τις πολίτες παρά να τους φέρνουμε κοντά στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένουμε ε, στο να γίνεται δημόσια ακρόαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ τίθεται το ερώτημα, εμείς οι ίδιοι ως Επιτροπή Αναφορών μπορούμε να παίξουμε ε, κάποιο σημαντικό ρόλο. Η Νταϊάννα Γόλης και εγώ είμαστε στεναρά υπέρ αυτής της απόφασης ή αυτής της άποψης που λέει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι η κατεξοχήν επιτροπή που έρχεται σε επαφή με τους πολίτες. Γι' αυτό είπαμε στο γράμμα μας ότι το Κοινοβούλιο ε, μέσω της αρμόδιας επιτροπής ανα πάσα στιγμή μπορεί να συμμετέχει, να κάνει δικές του ακροάσεις, ανα πάσα στιγμή της διαδικασίας, καθ' όλη τη διάρκεια της συλλογή των υπογραφών. Αλλά και στην τελική ακρόαση αυτή να γίνεται κοινή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ε, το, την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Αυτά είναι για μένα τα σημαντικότερα σημεία στο σχέδιό μας και μέλημά μας να τα παρουσιάσουμε όσο γίνεται πιο ε, σαφώς Να σας πούμε τι θέλουμε εμείς λοιπόν. Και την άλλη φορά να συζητήσουμε και κείμενο. Για να δούμε και ποιες είναι οι ειδικές απόψεις και να τις συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ευχαριστώ συνάδελφε Χέφνερ. Μας δώσανε πέντε λεπτά οι διερμηνείς, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ. Αλλά για να συνεχίσουμε, αν θέλετε να συνεχίσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Λοιπόν, πρόκειται για μια συνενετική σιωπή.